Συνάδελφοι, καλημέρα Και χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφέρετε να βρείτε το δρόμο σας, να έρθετε εδώ και ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες γιατί σε όλες τις περιοχές ε, της Ευρώπης ε, που πολλές φορές δεν έχουν και εμπειρία με το χιόνι Υπάρχουν προβλήματα, κάποιες αεροπορικές εταιρείε δεν πετάνε. Από την Ισπανία έχουμε και άλλες δυσκολίες, όχι μόνο χιόνι, καταλαβαίνετε. Και επιπρόσθετα, στις 2.30 ξεκίνησε ο τρομερής διάλογος. Άλλος ένας τρομερής διάλογος δηλαδή. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν ε, στον τρίλογο, στον τριμερή αυτό διάλογο. Η κυρία Τρούπελ, η Συντόνια, ο κύριος Μπούγκε, Γέντζεν, Φέρμ. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κύριος Στέφαν Λέναρτ δεν μπορεί να έρθει, αλλά είναι πολύ εγωιτευτική η κυρία που τον αντικαθιστά. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε πια τίποτε ευθύνη για τον τριμερή αυτό διάλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να ε, αντιδράσουμε με μια κάποια ευελιξία. Επειδή και η μερίσια διάταξη είναι τέτοια, που πραγματικά πρέπει να συζητηθεί με το σωστό και δέοντα τρόπο. Προκειμένου με τον τρόπο αυτό, να ολοκληρωθούν και οι οριζόντιες συζητήσεις μας ή εν πάση περιπτώσει να πάρουν ένα προσωρινό τέλος. Έχετε λοιπόν την ημερήσια διάταξη, την έχετε πάρει και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις. Για να ρίξω μια μάτια, δεν βλέπω κανέναν να είναι αντίθετος. Αποφασίζεται λοιπόν η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Όπως σας είπα, όπως σας έχω πει, πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της ε, ομάδας, της φάσης μάλλον περισυλλογής. Δηλαδή μετά από τη σημερινή συνεδρίαση όπου θα συζητήσουμε τα οριζόντια θέματα και θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, θα ακολουθήσει η κατάρτιση εγγράφων εργασίας, τα οποία θα τα καταρτήσει ο εισηγητή μας και βάση θα αποτελέσουν τα έγγραφα προσύλλογης όπως τα έχουμε συμφωνήσει και αυτά τα working documents, αυτά τα έγγραφα εργασίας, τα οποία θα τα καταρτήσει ο εισηγητής πριν από τα Χριστούγεννα, πριν από τις διακοπές θα αποτελέσουν απόρρια των εγγράφων περισυλλογής, των διαφόρων συζητήσεων και των ε, εισηγήσεων των συναδέλφων. Ο εισηγητής, λοιπόν, θα μας ε, υποβάλει κάποια έγγραφα εργασίας, όλα στα αγγλικά και πριν ε, τις διακοπές των Χριστουγέννων, μέσα στο 2010 δηλαδή, για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για τη στρατηγική για το 2020 της Ευρώπης και το έγγραφο εργασίας που θα αποτυπώνει όλα όσα θα συζητήσουμε εδώ σήμερα σε ό,τι αφορά την ε, διάθρωση, τη διάρκεια, τη διάρκεια και την ευελιξία του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, των δημοσιονομικών προπτικών. Και επίσης ο εισηγητής ανέφερε ότι έχει και ένα έγγραφο εργασίας για την εφαρμογή και την χρηματοοικονομική διαχείριση εντός των δημοσιονομικών προοπτικών. Θα μας υποβάλει λοιπόν και το έγγραφο αυτό. Και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Κυρίως για όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ε, υποβάλει τις προτάσεις, τις προτάσεις της για την απλοποίηση. Η Ιανουάριο του 2011 το περιμένουμε αυτό. Και αυτό λοιπόν θα ενταχθεί στον πλαίσιο των οριζόντιων θεμάτων, στη φάση της περισυλλογής. Αλλά ασφαλώς χρειαζόμαστε και την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρωτού μπορέσουμε και εμείς να δημοσιοποιήσουμε το έγγραφο εργασίας μας. Τον Ιανουάριο τώρα, την πρώτη εβδομάδα των εργασιών, όλα αυτά τα έγγραφα εργασίας θα έχουν ήδη μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Θα έχουν δημοσιευθεί πριν από τα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων θα έχουμε την ευκαιρία να τα εξετάσουμε στα αγγλικά και τον Ιανουάριο πλέον θα τα λάβουμε σε όλες τις γλώσσες, μεταφρασμένα. Σε περίπτωση τώρα που άλλοι συνάδελφοι από άλλες επιτροπές μας ζητήσουν τα έγγραφα εργασίας να δημοσιευτούν και στην ιστοσελίδα μας, εμείς έχουμε συμφωνήσει τα έγγραφα αυτά περί να είναι έγγραφα εργασία για μας. Και μετά όμως, στη συνέχεια δηλαδή, τα έγγραφα εργασία τα οποία θα έχει καταρτήσει πλέον ο εισηγητής, να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας. Στην αρχική μας σελίδα. Προκειμένου να μπορούν να τα επισκεφτούν και οι συνάδελφοι από τις άλλες επιτροπές σε περίπτωση που το επιθυμούν. Γι' αυτό λοιπόν Ξέρω φυσικά ότι όλα αυτά συζητιόνται και είναι λίγο αμφιλεγόμενα και στις άλλες επιτροπές, αλλά τα αποφασίσαμε αυτό γιατί είπαμε ότι τα έγγραφα εργασίας ουσιαστικά αποτυπώνουν τις σκέψεις μας. Εξακολουθούν φυσικά να είναι έγγραφα του εισήγητη, αλλά θέλουμε να συμπεριληφθούν τα στοιχεία της συζήτησης από πλευράς του εισηγητή και γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ πιο ευρεία η βάση από ό,τι στα έγγραφα περισυλλογής και οι επιτροπές που θέλουν να ασχοληθούν με το έργο μας θα έχουν έτσι μια επισκόπηση του τι συζητιέται εδώ στην Επιτροπή μας. Στους συντονιστές τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, συζητήσαμε το σχέδιο εργασίας για το επόμενο έτος και το ψηφίσαμε. Έγιναν κάποιες μικρές τροπολογίες, κάποιες μικρές αλλαγές. Νομίζω ότι πλέον όλοι έχετε το έγγραφο αυτό στην διάθεσή σας και οι συνάδελφοι εκείνοι που θέλουν να το διαβιβάσουν στις επιτροπές της άλλες. Μπορούν να σημειώσουν ποιο θέμα θα συζητηθεί σε ποια, και ποια, σε ποια ημέρα. Σε κάθε ημέρα. Και φαντάζομαι ότι κάποια θέματα θα απασχολήσουν και θα προσελκύσουν και συναδέλφους από τις άλλες επιτροπές. Επίσης, τι άλλο κάναμε. την τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών είπαμε ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε μια επιπλέον συνεδρίαση. Να τη βάλουμε κάπου στο πρόγραμμά μας προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα εκείνα τα οποία δεν καλύπτονται ακόμη από το πρόγραμμα εργασίας μας. Δεν έχουμε βρει κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά στη φάση των τομεακών θεμάτων θα ενταχθεί και αυτή η ημέρα 25 Ιανουαρίου, 1η Φεβρουαρίου ίσως αν ε, έχετε κάποια παρατήρηση ή αν θέλετε να σημειώσετε τις ημερομηνίε αυτές με ένα ερωτηματικό για μια επιπλέον συνάντηση, συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Και εγώ την επόμενη εβδομάδα στο Τρασβούργο θα προτείνω στην ε, συνεδρίαση των ε, Προέδρων των Επιτροπών ότι είχαμε το θέμα αυτό γιατί ένα θέμα συνέπεσε και με την ε, συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Εγώ θα εκφράσω ότι είμαστε πρόθυμοι, εγώ και ο εισηγητής, να κοιτάξουμε τι γίνεται στις επιτροπές, όπως κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Μεταφορών, όπως το κάνουμε και σε αυτή την εβδομάδα, σε ό,τι αφορά την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά αν κάποιος έχει πραγματικά κάποια συγκεκριμένη ε, ανάγκη, κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, να μα το πει και θα κοιτάξουμε το χρονοδιάγραμμά μα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι φυσικά όλε οι γνωμοδοτήσει και όλε οι επιστολέ είναι ευπρόσδεκτε. αρκεί όμω να μας στείλετε εγκαίρω. Γιατί τέτοιε γνωμοδοτήσει, επιστολέ, υποδείξει οι οποίε καταφθάνουν υπερβολικά αργά, δεν μπορούμε να τις ε, πραγματευτούμε. Και θα ήθελα να σας το πω ξεκάθαρα αυτό και γι' αυτό λοιπόν αυτό και στις άλλες επιτροπές ε, να το τονίζετε ότι είναι σημαντικό οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών να φτάνουν τη σωστή χρονική στιγμή και όχι υπερβολικά καθυστερημένα. Πέραν τούτων, συζητήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών πώς θα είναι η... πώς θα διαμορφωθούν οι συζητήσεις μας και κατά πόσον θα θέλαμε να καλέσουμε τους αρμόδιους επιτρόπους και να συζητήσουμε μαζί τους ή κατά πόσον θα θέλαμε να καλέσουμε ε, εμπειρογνώμονες ή και μέλη των αρμόδιων επιτροπών κατά περίπτωση γιατί έχουμε πολλές ε, ε, γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας και τους αντίστοιχους εισηγητές αλλά και σκιώδες εισηγητές σε πολλές περιπτώσεις ή και δύο εισηγητές. Αποφασίσαμε όμως να μην είναι επίσημη αυτή η διαδικασία, γιατί πολύ απλά εμείς ως Επιτροπή θέλουμε να καθορίζουμε εμείς προς τα που θέλουμε να κινηθούμε και τι δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα θέλαμε να αφιερώσουμε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα σε τέτοιε δηλώσει, σε τέτοιε εισηγήσει. Άρα αποφασίσαμε λοιπόν να μην πέρα από την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην προσκαλέσουμε άλλους επιτρόπους γιατί τι έχουν να μας πούν πέρα από αυτά που αναφέρονται και στις ανακοινώσεις τους. Και τις ανακοινώσεις τις διαβάζουμε και μόνες, μόνοι μας. Δεν έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν μας φάνηκε πιο σημαντικό εμείς να συνειδητοποιήσουμε και να αντιληφθούμε ποια θέματα θέλουμε να προωθήσουμε και πώς εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα ζητήματα. Ωραία λοιπόν. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να περάσουμε στο 3 της ημερήσιας διάταξης. Βάσει λοιπόν του εγγράφου περισυλλογής του Σαλβαδόρ, του εισηγητή, θα συζητήσουμε τη διάρκεια του μεσοπρόθεσμου πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι συνάδελφοι ήρθαν εδώ πέρα στην Επιτροπή μόνο και μόνο για να συζητήσουν θέματα διάρκειας, τη διάρκειας του πλαισίου. Ωραία, λοιπόν, Σαλπαντρό, σου δίνει το λόγο για να κάνει την εισαγωγή. Muchas ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα στην Επιτροπή μας θα ασχοληθούμε με τη διάρκεια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Αλλά φυσικά οι περισσότεροι από εμά ε, περιμένουμε την έκβαση των διαπραγματεύσεων που γίνεται στις διπλανές αίθουσες για το προπολογισμό του 2011. Και θα εξαρτηθούμε φυσικά από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο διμερή διάλογο και από την έκβαση αυτής της ε, Επιτροπής. Εμείς με βάση το πρόγραμμά μας είχαμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με το καθόδε ζήτημα της διάρκειας του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα, αρχίσουν, ε, που αρχίσει να ισχύει ε, από το 2014. Έχετε λάβει το σχέδιο για τις δημοσιονομικές προοπτικές που είναι ένα είδος συμφώνου μεταξύ δημοσιονομικής ε, ειρήνης και σταθερότητας αφενός και ελαστικότητας αφετέρως προς τη χρήση των πόρων. Κανονικά μέχρι στιγμής οι δημοσιονομικές προπτυρικές στις τέσσερις περιόδους ισχύω τους διαρκούσαν μέχρι, από 5 μέχρι 7 χρόνια. πρώτη, το πρώτο απολύτες πλαίσιο ήταν 5 ετές. Αλλά το 1993 και μετά, όπως βλέπετε, η διάρκεια αυτού του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου ήταν ετής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμενε να καθένα ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να παρακολουθεί τους θεσμικούς ρυθμούς, να είναι συναφές με τους θεσμικούς ρυθμούς και στο μέτρο του δυνατού να συνέπιπταν οι εντολές, η διάρκεια εντολών Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και Επιτροπής με τη διάρκεια του πολιτούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου για λόγους διαφάνειας. Έτσι, στις 17 Μαΐου του 2006 το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα στο οποίο ζητούσαμε πενταετή διάρκεια για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ακριβώς για να συμπίπτει τη διάρκεια αυτού του πλαισίου με τις εντολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μπορούμε να έχουμε σταδιακά μια διαδικασία ε, facing in. Στην περίοδο όμως 2007-2013, στο ισχύον δηλαδή πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, στις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, παρόλο που είχαμε ψηφίσει να διατηρηθεί η πενταετία, για αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές προτιμήσαμε την επταετία. Για την, για την πολιτική συνοχή και για την περίοδο της κοινή γεωργικής πολιτικής ήταν σκόπιμο να έχουμε ένα διαρκέστερο δημοσιονομικό πλαίσιο για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων και την πλήρη εκτέλεση και εφαρμογή των ε, διαρθρωτικών πολιτικών και της γεωργικής πολιτικής. Για τις επόμενες όμως δημοσιονομικές προοπτικές, που είναι αντικείμενο της δικής μας εντολής, Επιτροπής ε, ΣΟΥΡ, θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ σταθερότητας αφενός και ελαστικότητας αφετέρου. Γιατί θα ζήσουμε σε μια περίοδο με πολύ ισχνούς δημοσιονομικούς πόρους ε, που όλα θα γίνονται με σύνθημα τη λιτότητα. Οπότε η διάρκεια και των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών θα είναι ένα ακόμη στοιχείο για να ενισχυθεί η ελαστικότητα του κοινοτικού προϋπολογισμού. η πενταετής διάρκεια, αυτό ο πενταετή κύκλο θα μα εξασφαλίσει έναν απόλυτο παραλληλισμό και σύμπτωση μεταξύ τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών και τη διάρκεια τη εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή. Βέβαια, θα χρειαστεί και η θέσπιση μιας περίοδου σταδιακή εισαγωγή, ενό facing in, ώστε να συμπέσουν οι δημοσιονομικέ προοπτικέ με τι εντολέ και τι διάρκειε ε, εντολών του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή πριν να εξετάσουμε τις αναλλακτικέ λύσεις, θα ήθελα να σας πω ότι δημοσιονομικές προοπτικές που θα ξεπερνούν την πενταετία θα απαιτούσαν μια πολύ ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης. Μια ρήτρα που θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως στη Διοργανική Συμφωνία και στον κανονισμό για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ακόμη δεν έχουμε τον προϋπολογισμό του 2011 γιατί δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και να αποκαταστήσουμε μια γνήσια ε, σχέση εμπιστοσύνης ό,τι αφορά τη χρήση της ελαστικότητας και της ε, ρήτρα αναθεώρησης. Είναι παρακινδυνευμένο να πούμε σήμερα ότι μια πιο παρατεταμένη περίοδος ε, πέραν της πενταετίας δηλαδή με μια ρήτρα, αυστηρή ρήτρα αναθεώρηση θα γινόταν αποδεκτή από το Συμβούλιο. Οι εναλλακτικέ λύσει περιλαμβάνονται στη, σελίδα 4 του εγγράφου. Έχουμε την πρώτη ε, πρόταση που ξεκινάει με πενταετή δημοσιονομικέ προοπτικέ που θα ξεκινά το 2014. Δεύτερη εναλλακτική λύση είναι πάλι πενταετή ε, διάρκεια, αλλά που θα αρχίζει το 2021. Μετά από μια μεταβατική περίοδο πάλι επτάετη για τις δημοσιονομικές προοπτικές του 2014-2020 ώστε να πετύχουμε απόλυτο συγχρονισμό των εντολών του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Μία τρίτη εναλλακτική λύση είναι και πάλι πενταετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ξεκινά όμως το 2016 μετά από μία παράταση και προσαρμογή των υφισταμένων δημοσιονομικών προοπτικών και η τέταρτη εναλλακτική λύση, η λύση 4, είναι αυτή που εξετάζει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα δεκαετές πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με μια ρητή και ισχυρή ρήτρα ενδιάμεσης αναθεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλεί τη ρήτρα αυτή 5 συν 5. Κατόπιν στο έγγραφο αυτό του προβληματισμού έχετε και ένα σχεδιάγραμμα για να έχετε και μία οπτική απεικόνηση αυτών των προτάσεων με τις εντολές του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής με τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών και νομίζω ότι έτσι με την εικόνα αυτή έχουμε πολύ καλύτερες εξηγήσει. Τώρα, για να επισέλθουμε λίγο στις λεπτομέρειες. Η πρώτη πενταετής πρόταση που ξεκινάει το 2014, χωρίς το Facing In, μας δίνει την μέγιστη ελαστικότητα και είναι αυτή που εξασφαλίζει το μεγαλύτερο παραλληλισμό μεταξύ της εντολής του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της διάρκειας των δημοσιονομικών προοπτικών. Βέβαια, αυτή η πρώτη λύση, το πρώτο σενάριο, έχει κάποιες αδυναμίες. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να έχει κάποιο λόγο και ούτε θα βελτιωθεί η διαφάνεια και η δημοκρατική ευθύνη των θεσμικών οργάνων. Από πολιτική άποψη λοιπόν αυτή η πρώτη εναλλακτική λύση που έχει νόημα από τεχνική άποψη αν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ελαστικότητα, από πολιτική άποψη είναι ανέφικτη. Η δεύτερη εναλλακτική λύση κατά τη γνώμη μου είναι και πιο ενδιαφέρουσα προβλέπει πενταετής δημοσιονομικές προοπτικές που θα ξεκινούν από το 2021 με μια σταδιακή εισαγωγή, ένα facing in, μετά από μια επταετή μεταβατική περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Η δεύτερη αυτή εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι και πιο ενδιαφέρουσα, ενέχει όμως το πρόβλημα ότι ε, το επόμενο κοινοβούλιο δεν θα έχει την ευκαιρία διαπραγμάτευσης για τις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά ούτε και για τις επόμενες. Βέβαια αυτή η δεύτερη εναλλακτική λύση επιτρέπει στο μέλλον το 2021 μία απόλυτη ευθυγράμμιση και σύμπτωση των εντολών ε, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Οπότε από πολιτική άποψη είναι ενδιαφέρουσα αυτή η εναλλακτική λύση και φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα. Η τρίτη εναλλακτική λύση είναι αρκετά ελκυστική, μια και τώρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές μεταξύ των κρατών μελών. Προβλέπει πενταετή διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ξεκινώντας από το 2016 μετά από μια παράταση και προσαρμογή των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών. Η ρήτρα αυτή, ή μάλλον η εναλλακτική λύση αυτή έχει κάποια προβλήματα για το Κοινοβούλιο, όχι πολιτική υφή, αλλά περισσότερο τεχνική γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει πρόβλημα, γιατί η, παράταση, η πρόταση παράταση θα γίνει από την Ενενεργή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει καμία δυνατότητα γνωμοδότης ως προς τις δημοσιονομικές προοπτικές που θα αρχίζουν το 2016. Οπότε, από αυτή την άποψη, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τρίτη εναλλακτική λύση δεν είναι τόσο ελκυστική. Πάντως, και η εναλλακτική αυτή λύση σε περίπτωση μπλοκαρίσματος με το Συμβούλιο για τις δημοσιονομικές προοπτικές δίνει μια λύση. Την περασμένη φορά είχαμε την Αγγλική, Λουξεβουριανή και Αυστριακή Προεδρία. Τρεις δηλαδή διαδοχικές προεδρίες χρειάστηκαν για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές την τελευταία στιγμή. Οπότε, δεδομένης της ε, κατάστασης, ε, της δινής δημοσιονομικής κατάστασης και της λιτότητας, Ίσως τα δύο χρόνια 2011 και 2012 δεν είναι η καλύτερη περίοδος για διαπραγμάτευση πλήρων δημοσιονομικών προοπτικών. Οπότε ίσως η πρόταση για την παράταση των ισχυωσών ε, δημοσιονομικών προοπτικών δεν είναι κακή. Και έχουμε και την τέταρτη εναλλακτική λίστα της δεκαετής δημοσιονομικές προοπτικές με ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης 5 5. Με βάση τα ανώτατα όρια με, όλο, με όλους τους μηχανισμούς και τα νομικά μέσα αλλά και με τις πολιτικές συνοχής γεωργίας και των διαφορετικών πολιτικών είναι σημαντική αυτή η επιλογή αλλά χρειάζεται απαραίτητη ελαστικότητα για να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτής της ρήτρας ενδιάμεση αναθεώρησης. Πάντως μέχρι τώρα η εμπειρία που είχαμε από την ενδιάμεση αναθεώρηση δεν μας γεμίζει και με αισιοδοξία για να επικροτήσουμε την τελευταία αναλλακτική λύση του δεκαετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχει κάποια πλεονεκτήματα αυτή η λύση 4, αλλά έχει και μειονεκτήματα γιατί προσδιορίζει και παγιώνει όλες, όλα τα ανατοτόρια δαπανών, άρα μαστερεί την ελαστικότητα. Επίσης, η Κομισιόν προτείνει αποθεματικά σε όλες τις κατηγορίες. Είναι προφανέ βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να, εξα... να εξακριβώσουμε κατά πόσο το Συμβούλιο για τα κράτη-μέλη θα ήταν πρόθυμα να προβλέψουν σημαντικά αποθεματικά υπερηθόρια σε όλες τις κατηγορίες δαπανών. Αυτό μου φαίνεται αρκετά περίπλοκο το σημερινό Συμβούλιο να δεχτεί μια τέτοια πρόταση. Και στο τέλος του εγγράφου περιλαμβάνω κάποιες ερωτήσεις που είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν. Η πιο σημαντική ερώτηση είναι πώς θα συνδυάσουμε την ελαστικότητα με την ανάγκη να έχουμε αρκετά μακροχρόνιους κύκλους προγραμμάτων, ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχή και στη γεωργική πολιτική. Πώς θα συγχρονίσουμε στο μέλλον αυτά τα πολιετή προγράμματα με τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Και άλλες δύο ερωτήσεις στο τέλος του εγγράφου. Από στρατηγική άποψη, ποια είναι η καλύτερη λύση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, οποίες το Κοινοβούλιο ευελπιστεί ότι θα συμπεριλαμβάνεται, γιατί αυτή είναι μία από τις ελίτες που εξετάζει σήμερα ο τριμερής διάλογος, Οπότε θα τα σκόπιμο να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές το 2011 ή να διαπραγματευτούμε μια παράταση των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών δεδομένου του δημοσιονομικού και του πολιτικού πλαισίου στις διάφορες χώρες μέλη της Ένωσης. Και η τελευταία ερώτηση είναι πιστεύετε ότι η ρήτρα 10 η τέταρτη εναλλακτική λύση απαιτεί μια υποχρεωτική ε, ρήτρα ενδιάμεση αναθεώρησης. Και πώς θα μπορούσε αυτό να ενταχθεί σε μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές είναι οι προκαταρκτικές ερωτήσεις που θέτω προς συζήτηση. Έχετε λάβει και ένα πίνακα από τη γραμματεία για να δείτε πώς απεικονίζονται αυτές οι τέσσερις εναλλακτικέ ε, λύσεις με υπό το πρίσμα τεσσάρων ε, σημαντικών ενιών όπως είναι η ελαστικότητα, η διαφάνεια των κοινοβουλευτικών και πολιτικών αποφάσεων, η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα στην διαχείριση των πολιτών προγραμμάτων και η σταδιακή εισαγωγή, το facing in, πώς συμπεριλαμβάνεται στις τέσσερις αυτές εναλλακτικές προτάσεις. Ελπίζω να σας προσανατολίσει κάπως αυτό το σχέδιο. Η πιο συνετή και λογική επιλογή από πλευρά Συμβουλίου θα ήταν να κρατήσουμε το σημερινό στατουκβό, το 7 ετές, μια και είχαμε τέσσερις διαδοχικές περιόδους δημοσιονομικών προοπτικών 7 ετής και η πλειοψηφία στο Συμβούλιο είναι υπέρ της επταετίας, της επταετούς διάρκειας του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό όμως είναι το στάτου Ακούω, οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση ή ανάλυση εκ μέρους μου. Είναι γνωστή αυτή η κατάσταση. Αυτά είναι η εισαγωγή, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Das war... Σας ευχαριστώ. Αυτά εισαγωγικά λοιπόν σε ό,τι αφορά το έγγραφο περισυλλογής το οποίο το είχατε στη διάθεσή σας από την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, είχατε στη διάθεσή σας το Σαββατοκύριακο να εξετάσετε τα διάφορα θέματα. Και τώρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί συνήθως θα είχαμε τον, ε, σε κανονικές συνθήκες θα είχαμε τον γύρο των συντονιστών. Αλλά λόγω του ότι έχουμε αυτή την ανταγωνιστική εκδήλωση του τριμερού ε, διαλόγου που γίνεται παράλληλα με, με την συνεδρίασή μας, δεν έχουμε ε, όλους τους συντονιστές. Δεν έχει το έλκτο συντονιστή του εδώ και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θα έχουν ρυθμίσει τα πράγματα. Θα αντικαθίσει ο Αίνταν τον ε, Γιώραν. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τους φιλελεύθερους, με τους πράσινους. Είναι εδώ πέρα και κάποιοι συνάδελφοι, το FND. Επίσης δεν ξέρω. Η FD. Για το ΕΛΚ. Ποιος θα μιλήσει. Ο κύριος Καράς. Ωραία λοιπόν. Και οι φιλελεύθεροι να το σκεφτούν. Εσείς κύριε Άλβαρο, α όχι, εντάξει. Ότμαρ λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι πρέπει να πούμε ότι ειλικρινά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ε, να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα από πλευράς ομάδας. Αλλά να σας πω εγώ εκ μέρους μας το εξής. Βρισκόμαστε σε μια επιτροπή η οποία δεν έχει μόνο καθήκον να προγραμματίσει τα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά έχουμε να κοιτάξουμε τις ειδικές ε, προκλήσεις ε, της πολιτικής και σε ό,τι αφορά το, τα δημοσιονομικές, ε, τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να διδαχτούμε από τα παθήματα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2011. Να μην είμαστε υπερβολικά τεχνικοί σε αυτή την προκαταρτική φάση και να μην, ε, προ... να μην προσανατολιζόμαστε ιδιαίτερα σε χρονικό πλαίσιο. Να μην κοιτάμε τόσο έντονα πόσο... πώς θα δράσουν τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να βρούμε, ε, αν θέλετε, ένα κοινό σημείο και να πείσουμε την δημόσια γνάμη πόσο απαραίτητες είναι αυτές οι δημοσιονομικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό λοιπόν θα κριθεί από το περιεχόμενο. Θα κριθεί από το πώς θα διαμορφωθεί ο προπολογισμό μέχρι το 2020. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις, όπως είπε ο εισηγητής, άσχετα από τις ε, από τον προγραμματισμό για ρήτρα αναθεωρήσεις και φυσικά τα θέματα ευελιξίας και διαφάνειας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και τα θέματα της ασφάλειας δικαίου. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τις δημοσιονομικές προοπτικές και να κοιτάξουμε μια αξιολόγηση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και να κοιτάξουμε με κριτικό τρόπο τα μέσα τα οποία δαπανήθηκαν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την έκταση του ελεκτικού συνεδρίου. Κατά δεύτερο, θα ήθελα να ζητήσω και να ρωτήσω κατά πόσο παίζουν ρόλο οι εμπειρίες μας από την κρίση, γιατί συνειδητοποίησαμε στην κρίση ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει λοιπόν η πιο πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προπολογισμό. Όλοι λέμε ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την πιο πολύ έρευνα, ανάπτυξη και την επιστήμη. Κατά πόσο λοιπόν. Πόσο θα πετύχουμε αυτή την περισσότερη Ευρώπη σε ό,τι αφορά α, τον συντονισμό. Τι σημαίνει Small Business Act, Single Market Act, Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκή Εξωτερική ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τι σημαίνει το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, τι συνεπάγονται όλα αυτά για τον προϋπολογισμό, αυτή η νέα κατανομή των αρμοδιοτήτων τι σημαίνει, πώς αποτυπώνεται. Μιλάμε για πολιτικούς τομείς οι οποίοι ως τώρα δεν αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό και η ασπίδα η προστασίας. Πώς επηρεάζει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ στην παρούσα φάση θα ήθελα να οριστούν οι πολιτικές προτεραιότητες. Να κοιτάξουμε ποια είναι τα απαραίτητα νομικά μέτρα γιατί δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας με τον εφιστάμενο προϋπολογισμό και θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε χρήματα για αυτά που μας χρειάζονται. Πρώτα θα πρέπει να συμφωνήσουμε τους στόχους μας και μετά να δούμε τι θα πρέπει να ζητήσουμε για τις δαπάνες. Σας ευχαριστώ. Σα Dank Σας ευχαριστώ και αυτό που είπατε προς το τέλος ήταν πολύ σημαντικό γιατί μας ε, καταδεικνύει με σαφήνεια ότι το Συμβούλιο επιμένει στην παλιά του θέση. Αίντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον Σαλβαδόρ για το έργο που επιτέλεσε, το έγγραφο που εκπώνησε και την ξεκάθαρη ανάλυση των τεσσάρων εναλλακτικών λύσεων. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Κάρας. Όταν αρχίσαμε να προγραμματίζουμε το έργο της Επιτροπής, είχαμε ζητήσει οι σοσιαλιστές αυτό το θέμα της διαρθρώσης, ε, της ε, ελαστικότητας, της διάρκειας, το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το τελευταίο πράγμα που θα απασχολούσε την Επιτροπή, γιατί περιμέναμε πρώτα απ' όλα ε, μία στρατηγική ανάλυση, γενική ανάλυση για το στόχο που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές που την ενδιαφέρουν. Γι' αυτό ζητήσαμε να αφήσουμε για το τέλος το θέμα της διάρκειας των δημοσιονομικών προοπτικών. Ο Σαλβαντόρ μας εξήγησε τα υπέρ και κατά των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Δεν πρόκειται να, να τα επαναλάβω. Ο εισηγητής μας είπε ότι η επταετία γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Είναι κάτι γνωστό. Θα ήθελα όμως το έγγραφο να λέμε δύο λόγια και για αυτή την εναλλακτική λύση, γιατί είναι αρκετά έγκυρη. Γιατί μέχρι στιγμής φαίνεται σαν να ασχολούμαστε μόνο με τις πενταετής προοπτικές. Αλλά πιστεύω ότι και η επταετία είναι μια διάρκεια που έχει αρκετού. οπαδού. Γιατί να μην πούμε δύο λόγια και γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει αποκρισταλωμένη γνώμη για το ποια λύση προτιμά. Ίσως θα πρέπει να συνδυάσουμε όλες αυτές τις προτάσεις για το δημοσιονομικό, για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Καταρχήν, όταν μιλούμε για δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. να μην αρχίζουμε εκ του μηδενό να κάνουμε τάβουλα ράζα σαν να μην είχε γίνει καμία προεργασία μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό είναι ένας προϋπολογισμός που δεν είναι δεδομένος ακόμη. Δεν χρειάζεται να έχουμε ε, να αφιερώσουμε δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία. Έχουμε ήδη βάσεις. Δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε όλα από την αρχή. Τώρα, ποια είναι η καλύτερη ε, από τις αναλλακτικέ λύσεις του Σαλβαδόρ. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία που να διακρίνεται ως η επικρατέστερη. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τις ε, επικρατέστερες συμβαστικές λύσεις, όπως θα βγουν από τη συζητήση στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η επικρατέστερη λύση είναι η πενταετής για να υπάρχει σύμπτωση της διάρκειας του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου με τις θητείες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Κάτι που εξασφαλίζει σύμπτωση, διαφάνεια, δημοκρατικό έλεγχο. Είναι λογικό οι εντολές να συμπίπτουν και οι διάρκειες να συμπίπτουν. Αυτό είναι ένα επιχείρημα υπέρ της πενταετίας. Άλλοι όμως ισχυρίζονται ότι η πενταετία είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για ορισμένα πολυετή προγράμματα που μπορεί να είναι αυτά των συγκοινωνιών, του Ταμείου Συνοχής, τα ερευνητικά προγράμματα, ακόμη και τα προγράμματα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Για ορισμένα προγράμματα που θα πρέπει να τα προσδιορίσουμε είναι πιο δόκιμη μια πιο παρατεταμένη περίοδος, επταετής ίσως. Αλλά αν μας βολεύει για τέτοια προγράμματα η επτέτεια, μπορεί να μας εξυπηρετεί και η δεκαετία για την σταθερή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Τώρα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε δημοσιονομικό πλαίσιο πενταετές με ε, δεκαετές πλαίσιο για ορισμένα προγράμματα. Περίπου αυτό προτείνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το 5 συν 5. Με υποχρεωτική ρήτρα ενδιάμεση αναθεώρηση. Αλλά στην ενδιάμεση αναθεώρηση δεν χρειάζεται να τα αναθεωρήσουμε όλα. Κάποια να μένουν σταθερά. Και όλοι όσοι ζητούν σταθερότητα, ή πενταετία ή δεκαετία, είναι λογικό να είναι υπέρ τη μερική αλλαγή. Οπότε είμαι το 5 συν 5, είμαι πενταετή ε, δημοσιονομικέ προοπτικέ συν δεκαετή ορισμένα, δεκαετή διάρκεια για ορισμένα προγράμματα και αυτό είναι σκόπιμο. Όπως είπε ο Σαλβαντόρο ότι χρειαζόμαστε μία ρήτρα υποχρεωτικής ενδιάμεσα αναθεώρηση. Γιατί είδαμε τι συνέβη με την προηγούμενη αναθεώρηση. Να μην μείνουν ε, επί ξύλου κρεμάμενες οι δημοσιονομικές προοπτικές, οι μετέωρες. Είναι μια νομική λεπτομέρεια, νομικοτεχνική, αλλά πολύ σημαντική θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτή την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Νομίζω ότι αυτή η εναλλακτική λύση είναι αυτή που συνδυάζει τις ε, επικρατέστερες θέσεις. Αλλά πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν αυτές οι νέες προοπτικές. Ε, εμένα το θέμα της ε, διετούς παράτασης είναι πολύ σκόπιμο. Το θεώρησε και ο Σαλβαντόρ, ελπιστικό και εγώ το ίδιο πιστεύω. Βέβαια το Συμβούλιο δεν είναι καμία διάθεση για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή και σίγουρα αν έχει διάθεση διαπραγμάτευση δεν είναι παρόμοια με τη δική μα για τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Οπότε η διετή παράταση των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών δεν θα ήταν κακή και θα εξασφαλίσει και μια σταθερότητα. Γιατί η προσέγγιση του Συμβουλίου νομίζω ότι είναι επιβλαβής για τα δικά μας συμφέροντα. Και μία άλλη, κατά τη γνώμη μου, θετική ιδέα που συνάδει υπέρ της παράτασης, της διετούς παράτασης των υφισταμένων προοπτικών είναι τα προβλήματα που είχαμε στα διαρθρωτικά προγράμματα. Στην αρχή του δημοσιονομικού πλαισίου είχαμε μια πολύ αργή κίνηση. Φαίνεται όμως ότι άρχισαν να δραστηριοποιούνται τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή, οπότε με τη διετή παράδοση των διαρθρωτικών ταμείων θα εξασφαλιστούν οι χώρες που εξαρτώνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και θα μπορέσουν ανυφάλια να προβούν στο, στην εφαρμογή και των υπόλοιπων προγραμμάτων. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Κύριε Άλβαρο για τους φιλελεύθερους τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να σας ε, κάνω μία μικρή πρόταση. Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα που μας προτείνει ο Σαλβαδόρ. Καταρχάς σας ευχαριστούμε για την ε, πρόταση αυτή, γιατί δεν είναι απλό να κάνει κανείς τέτοια, τέτοιες προτάσεις, γιατί κυρίως θα πρέπει να κοιτάξουμε και την εφικτό, όχι το τι θα ήταν μόνο θεμητό. Θα πρέπει ως κόκκινη γραμμή να κρατήσουμε αυτά που αφορούν τον δημοκρατικό έλεγχο, ότι υπάρχει δηλαδή ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο καθορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο και συμμετέχει στην εκτελεστική. Νομίζω ότι είναι καλή δημοκρατική παράδοση να μην λαμβάνονται αποφάσεις τις οποίες μετά ε, πρέπει να εκτελούν για παράδειγμα ένα νέο κοινοβούλιο. Γιατί αυτό θα συνέδινε υπέρ της πρώτης λύσης ε, να συνεχιστούν οι δημοσιονομικές προεπτοκές με το 2014, αλλά αυτό τι θα σήμαινε α, ότι θα υπήρχε αυτή η δημοσιονομική προοπτική 2014 και 2019, αλλά αυτό τι θα σήμαινε ότι οι συνάδελφοι μετά από εμάς που θα εκλεχθούν μετά δεν θα μπορούσαν να καθορίσουν και θα έπρεπε να εκτελέσουν μία απόφαση την οποία δεν έλαβαν οι ίδιοι. Ως εκ τούτου, για να μην κοιτάξουμε τι είναι δύσκολο να πραγματοποιήσουμε και για να είμαστε σύντομοι, θα ήθελα να περιοριστώ στο σημείο 3, τα οποία θεωρώ ότι είναι το πιο ρεαλιστικό, αλλά όχι με την απεριόριστη ικανοποίηση την οποία εξέφρασε η συνάδελφος των σοσιαλιστών, αλλά με κάποιε αμφισβητήσει. Καταρχά τα θετικά. Η λύση 3 προσφέρει για την δημοσιονομική προοπτική το 2016, τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ξεκινήσει το 2014 να κάνει τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Άρα να υπάρχει αυτή η σύνδεση που θέλουμε. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα το προτείνει αυτό το 2013 δεν είναι τόσο επιθεμητό γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαντάζομαι θα θέλει να έχει και αυτή μια συνέχεια. Και δεν μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Και θεωρώ λοιπόν ότι η λύση 3 από πλευράς ε, δημοκρατικού ελέγχου είναι η πιο σωστή να κάνει το Κοινοβούλιο την πρόταση αυτή το 2014. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε και γι' αυτό δεν είμαι τόσο απεριόριστα ικανοποιημένος όπως ο συνάδελφος είναι το εξής. Αν υπάρχει ε, παράταση της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδους, να δούμε από ποιους όρους θα γίνει αυτό, γιατί έχουμε και την ανταγωνιστική εκδήλωση που πραγματεύεται το θέμα αυτό και αν υπάρχει τέτοια παράταση δεν νομίζω ότι μπορούμε να εκδώσουμε μια λευκή επιταγή. Όχι, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι όροι, ότι θα πρέπει να λεφτούν υπόψη τα συμφέροντά μας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι όροι, ποιοι είναι οι συνθήκες, να μας πει ίσως ε, ο εισηγητής υπό ποιους όρους θα έγινε η παράταση αυτή. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν προβληματικό να ισχύει το πλαίσιο αυτό μόνο για πέντε χρόνια. Είναι λογικό μάλιστα γιατί είδαμε ότι στην τρέχουσα αλλά και στην τελευταία ε, θητεία άλλαξαν πάρα πολύ ε, γρήγορα και ραγδαία οι συνθήκες οι οποίες επιτάσσουν τελικά διαφορετική προσαρμογή και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι αν ε, επικεντρωθούμε στην ε, λύση 3 θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σαλβαντόρ για τη δουλειά του. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος και τώρα νομίζω Φρανσουά για τους πράσινους. Oui, Madame la Présidente. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή για ε, όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει. Είναι πάντοτε πολύ συνοπτικά και διαφωτιστικά τα όσα μας παρουσιάζει. Για την επιλογή 3 εγώ έχω μια επιφύλαξη όσον αφορά το πολιτικό χρονοδιάγραμμα. Γιατί το τεχνικό χρονοδιάγραμμα το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πού βασίζεται για να μας κάνει αυτές τις προτάσεις ο εισηγητής. Όμως από πολιτική άποψη θα είχαμε ακόμα δύο χρόνια ε, τις ίδιες δημοσιονομικές προοπτικές που ισχύουν πριν να υπάρξει η, η χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι λοιπόν αποδεκτό να περατείνουμε για δύο χρόνια προοπτικές τις οποίες είχαμε σκεφτεί και εγκρίνει ενώ δεν υπήρχε κρίση. Και έπειτα Επίσης δεν είχαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σήμερα δηλαδή έχουμε μια νέα ευθύνη για την επεξεργασία των προοπτικών και δεν θα ασκούσαμε αυτές τις νέες μας ε, αρμοδιότητες αν το κάναμε αυτό. Άρα λοιπόν στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα θα έλεγα ότι δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο και έπειτα για τη διάρκεια την, την πενταετή που λέτε ότι είναι καλό να συμπίπτουν οι περίοδοι προγραμματισμού με τις περιόδους θητείας αλλά Παρ' όλα αυτά, ο προγραμματισμός θα πρέπει καλύτερα να συνδυάζεται με το ρυθμό των πολιτικών και του προγραμματισμού. Και νομίζω ότι πενταετής προγραμματισμός είναι κάπως σύντομο. Ιδιαίτερα για την συνοχή, ο ρυθμός των 7 ετών πάλι πολλέ φορέ κρίνεται ε, σύντομο. Τώρα αν θα πρέπει να ξανάρθουμε στα 5 χρόνια, ξέρω ότι η Κομισιόν αυτό επιθυμεί, αλλά εγώ δεν είμαι πεπισμένος. Και, εν πάση περιπτώσει, περιμένω κάποια επιχειρήματα για να μα δείξει όντω ότι αυτό συμπίπτει με την πραγματικότητα επιτόπου. Τώρα, ίσως σε δύο χρόνια μπορεί να υπάρχει λιγότερη λιτότητα, άλλε κυβερνήσει θα διαπραγματευτούμε καλύτερα όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου. Αλλά ούτε και αυτό είναι βέβαιο. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα να πιάσουμε τον τάβρα από τα κέρατα και να επιβάλλουμε τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ώστε να μπούμε σε ένα προγραμματισμό και σας λέω αυτό τώρα προσωπικά ε, γιατί η ομάδα μου ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Νομίζω πάντως πως πιο ρεαλιστική επιλογή είναι οι δύο. Σας ευχαριστώ, Ρίτσαρντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ομάδα μας δεν είχε το χρόνο να συγκεντρωθεί και να το συζητήσει, άρα σας δίνω τη δική μου προσωπική άποψη. Και εγώ... Ε, ε, θα θεωρήσω ως ε, φυσιολογικό το επταετές πρόγραμμα που ισχύει αυτή τη στιγμή. Ε, ικανοποιεί την απέτηση για σταθερότητα που χρειαζόμαστε για το μακροχρόνιο προγραμματισμό όσον αφορά ας πούμε την συνοχή και την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα και γι' αυτό το λόγο υποψιάζομαι γίνεται η σημερινή συζήτηση. Καταρχήν λείπει δημοκρατικός έλεγχος το σύστημα του πολιετούς πλαισίου είναι μια έννοια που, εννοείται, που κατανοείται από την κοινή γνώμη ε, πολύ λίγο και νομίζω πως σίγουρα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό θέμα. Άρα ευθυγράμμιση καλύτερη με το εντολές τη θητεία του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν κατά την άποψή μου θα ήταν ε, ωφέλιμο και αυτό επιτυχάνεται περισσότερο με πενταετές πρόγραμμα. Έπειτα, δεύτερο ζήτημα αφορά την ευελιξία και όπως είπαν και διάφοροι ομιλητές, οι καιροί αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τη σήμερα ημέρα και γι' αυτό είναι πολύ, σημαντικό οι προτεραιότητες της Ένωσης να αναθεωρούνται διαρκώς και να υπάρχει μια διαδικασία μέσω της οποίας αυτό θα γίνεται σε τακτική βάση. Και δεν θεωρώ πως αυτό είναι αντιφατικό με το μακροχρόνιο προγραμματισμό της σταθερότητα και τους ε, κατηγορίες 1 και 2. Πιστεύω πως επίσης θα είναι πιο λιτή οι προϋπολογισμοί, τα περιθώρια θα είναι στενότερα και άρα η ευελιξία θα είναι πλονέκτημα. Εν κατακλείδη, εγώ είμαι υπέρ πενταετούς προγράμματος. Ε, πέντε συν πέντε αυτή η ιδέα με ενδιαφέρει από την Κομισιόν, αλλά αν αυτό σημαίνει ότι αυτή η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα είναι αρκετά στεναρή, ε, ίσως τότε θα έπρεπε να κάνουμε ένα τελείως καινούριο πενταετές πρόγραμμα. Αν όχι, ένα δεκαετές πρόγραμμα θα αυξήσει την πιθανότητα του να προκύψουν προβλήματα όπως αυτά που έχουμε τώρα και αυτό είναι βλαβερό για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ του πενταετούς προγράμματος εγώ και, και βρίσκω και, και σύμφωνος με τον τρόπο που γίνεται το phase-in. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μιγγέλ Πόρτας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πρώτη παρατήρηση για το χρόνο και για την οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι όταν συζητάμε αν ο προγραμματισμός θα πρέπει να είναι πενταετής ή επταετής, θα πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι σημαίνει και σε τι έχει μετατραπεί αυτός ο προγραμματισμός για τον οποίο συζητάμε και κατά πόσο αυτό αποτελεί μια ε, άσκηση εξουσίας και σύγκρουση δυνάμεων τελικά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν στον προϋπολογισμό, όμως ε, δεν πρόκειται για έναν προγραμματισμό ε, δυναμικό, δεν πρόκειται για έναν δημόσιο προϋπολογισμό, για μια οικονομία που διαρκώς βλέπει αυξήσεις. αυτό που βλέπουμε, που διαπιστώνουμε στην ουσία, είναι μια αύξηση των ε, στιγμών αβεβαιότητας και γι' αυτό από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι ο πταετής προγραμματισμός τίνει να είναι σχεδόν πάντοτε κακή λύση. Σε αντίθεση ενός προγραμματισμού 5 συν 5 για το λόγο που ήδη αναφέρθηκε, ότι δεν υπάρχει δηλαδή καμία εγγύηση για μια σοβαρή αναθεώρηση στη ε, μέση της διαδικασίας. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε κάτι άλλο θα γίνει. Και είναι προφανές ότι 5 5 στην ουσία τίνει να μετατρέπει μια, σε μια απλή παράταση την δεύτερη πενταετία. Άρα λοιπόν αυξάνεται η ακαμψία του προγραμματισμού, ενώ αντιθέτως η οικονομία κάθε φορά φαίνεται να είναι όλο και πιο αβέβαιη. Πέρα από αυτή την ε, παρατήρηση, όταν θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα το πενταετές, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ξεκινήσει από το 2016. Ε, Για λόγους ε, πολιτικής φύσης Δηλαδή, το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λόγο που να μην, να μην είναι απλώς μια συνυπογραφή των όσων θα είναι οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Εμείς θα πρέπει να ε, λύσουμε τα προβλήματα δημοκρατικά στην Ευρώπη, το θέμα της χρήσης του προϋπολογισμού, γιατί Διαφορετικά, οι ευρωεκλογέ θα μείνουν και πάλι χωρίς μεγάλη συμμετοχή. Πιστεύω λοιπόν πως αυτή η Επιτροπή ΣΟΥΡ θα πρέπει να καταλήξει στο ανάγκη προστασίας των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών από τον κίνδυνο τις μηδενικής βάσεις για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Δηλαδή θα πρέπει περισσότερο να μιλήσουμε για συνέχιση των κατηγοριών που ήδη υπάρχουν στην, στον προπολογισμό. Και αμφιβάλλω πως θα το καταφέρουμε αυτό μέχρι το 2014. Έτσι όπως βλέπω τις πολιτικές σχέσεις που επικρατούν σε επίπεδο κυβερνήσεων. Και τελευταία μου παρατήρηση. Και νομίζω κάποιος σοσιαλιστής συνάδελφος το είπε αυτό, ότι δηλαδή ένα έτος διαπραγματεύσεων είναι υπεραρκετό. Και όσον αφορά την ευελιξία, πιστεύω πως θα πρέπει να είναι πιο ισχυρή από ό,τι τώρα, δηλαδή να είναι εντός των περιθωρίων του προϋπολογισμού, ε, μάλλον είτε είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού, είτε εκτός των ορίων του προϋπολογισμού. Υπέρ λοιπόν της πενταετίας ανάγκη να υπάρχει μεσοπρόθεσμη σταθερότητα για τις πολιτικές είτε είναι αυτές οι γεωργικές είτε είναι αυτές που συνδέονται με τα διευθυντικά ταμεία. Γιατί δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο όλα αυτά. Θα πρέπει να βασιστούμε σε μια καμπύλη που αρχίζει την ε, πρώτη χρονιά του δημοσιονομικού πλαισίου κατεβαίνει και μετά ξανανεβαίνει προς το τέλος του δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει δηλαδή να προβλέψουμε και μία, ένα ποσοστό των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών για προγράμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προβλεφθεί από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Ähm, Σας ευχαριστώ και να σημειώσω ότι και εγώ θεωρώ ότι μία μονοετής φάση διαπραγμάτευσης θα πρέπει να αρκέσει. Ωστόσο, προτού, προτού το σκεφτούμε αυτό καν, θα πρέπει με το Συμβούλιο να διαπραγματευτούμε και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα για να δούμε τελικά το πώς θα θέλουμε να καθορίσουμε την, ε, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά βλέπουμε ότι στην παρούσα φάση το Συμβούλιο αρνείται να διαπραγματευτεί μαζί μας και αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε διαρθρωτικά ότι και το Συμβούλιο χρειάζεται μόνο ένα έτος για να συμφωνήσει μαζί μας, τα πράγματα δυσκολεύουν. Τώρα από το EFD είναι κανείς εδώ. Να δούμε λοιπόν τώρα τους εισηγητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Engel Ellis, Marinescu, Reimers, Dantin, Ugias, Gönsch, ja, um, um, um... Uta, Uta, é só uma coisa. A opinião que eu dei, a opinião que... Uta ή να διευκρινίσω κάτι, ότι η γνώμη μου ήταν τελείως προσωπική, δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα στην ομάδα. Ναι, αλλά είμαι βέβαια ότι μπορεί να πείσει και του υπόλοιπου στην ομάδα σου. Άρα αυτή θα είναι η θέση τη ομάδα σου. Ωραία, λοιπόν. Η κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ, Γιούτα, και ελπίζω τα πράγματα να μην γίνουν όπως είπες και να το σκεφτεί η ομάδα. Ίσως να μην σας προκαλέσει έκπληξη το γεγονός γιατί είμαι από το 91 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την αρχή ασχολούμαι με την περιφερειακή πολιτική. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ασχολούμαι με δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα... Θα ήθελα μάλλον να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Γκαρίγκα για τις τέσσερις λύσεις που μας έδωσε, αλλά θα ήθελα να συμπεριληφθεί και μία επταετής ε, εναλλακτική λύση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι είδα φυσικά και οι βουλευτές ασχολούνται με δημοκρατικά θέματα και αυτόματα καταλήγουμε σε θέματα θητείας και σκεφτόμαστε με βάση τη θητεία. Αλλά η πολιτική συνοχή στην Επιτροπή αυτή ε, έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω να σκεφτείτε λίγο πώς σκέφτονται και οι πολίτες, να μπείτε λίγο στο μυαλό και των περιφερειών. Τι γίνεται όταν μιλάμε για πενταετή ή για επταετή ε, προοπτική. Ίσως να τα υπερβάλλω και λίγο. Θα ήταν καλό να διαπραγματευόμασταν για ένα έτος, αλλά δεν νομίζω ότι θα το ζήσω εγώ αυτό. Τα θεσμικά όργανα μπορεί να κάνουν διαπραγματεύσεις επί 2,5-3 έτη τα οποία, για θέματα τα οποία τελικά σε μία νύχτα και σε πολύ ομιχλώδες οποίο ε, αποφασίζονται και πάντα εις βάρος των περιφερειών, οι οποίοι τελικά ταλούζονται. και αν χρειαστεί τελικά να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα και να υπάρξει μια σύμπτυξη κατά 5 ή 7 έτη, εκεί θα έχουν προβλήματα, γιατί μετά τις διαπραγματεύσεις των 2,5 ετών θα πρέπει να κάτσουν να κοιτάξουν πώς μπορούν όλα αυτά τα σχέδια να μεταφραστούν σε καλά project, σε καλά σχέδια προς όφελος των περιφερειών και πώς μπορούμε να καταφέρουμε οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να επιτευχθούν στις διάφορες περιφέρειες και θα πρέπει να τονίσουμε και να τις αφηνίσουμε ότι αφενός τα δυόμιση έτη διαπραγματεύσεις και πέντε χρόνια ε, δημοσιονομικού πλησίου δεν αξίζουν τον κόπο. Θα πρέπει δηλαδή όλη αυτή η δέσμευση να αφορά μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο και κατά δεύτερον κοιτώντα τα διάφορα σχέδια δεν ολοκληρώνονται τα project αυτό σε δύο-τρία χρόνια. Μιλάμε για μακροπρόθεσμες, στρατηγικές, οικονομικές, οι οποίες προγραμματίζονται για, την, ε, για τις περιφέρειες και οι οποίες προϋποθέτουν πολύ απλά μια μακροπρόθεσμη χρηματική βεβαιότητα, όχι μόνο πέντε χρόνια. Και ακούγοντας το 2 επί 5 ή τα 10 χρόνια, θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτή η λύση μου φαίνεται ότι δεν έχει αρκετή ευελιξία, γιατί αν ε, χρειαζόμαστε μια καλή αναθεώρηση, δεν χρειαζόμαστε τα 10 έτη, μας φτάνουν τα 5 έτη και αν πούμε εκ των προτέρων ότι με την αναθεώρηση θα γίνει αυτό που γίνεται σήμερα και τελικά θα καταλήξουμε στα 10 έτη, πραγματικά πιστεύω ότι εκεί πέρα θα είναι αρκετά μη ευέλικτη κατάσταση, αρκετά άκαμπτη. Θα πρέπει να εξετάσουμε, θεωρώ, τις δημοσιονομικές προοπτικές 7 ετών. Και εγώ θεωρώ ότι έχει αποδείξει την αξία της αυτή η λύση. Κοιτώντας τον ίσιν 2, ίσιν 3 που θα προσθεθεί, το οποίο προϋποθέτει και μια σωστή αξιολόγηση μετά την ε, ολοκλήρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, θεωρώ ότι είναι καλύτερη λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα συμμετέχει στην ε, αξιολόγηση, στην κατάρτιση του δημοσιονομικού πλαισίου και ενδεχομένως για την τροποποίηση του προϋπολογισμού με κάποιους όρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευελιξία και στην τρέχουσα ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται κάτι τέτοιο, προβλέπεται ένα απόθεμα αλλά πρέπει να πω ότι οι εμπειρίες από τις τελευταίες ε, τρεις δημοσιονομικές προοπτικές κατέδειξαν για την πολιτική συνοχής ότι μπορούμε μεν να καταρτίζουμε στρατηγικές και σχέδια και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και προσθήκες, αλλά ότι θα πρέπει κυρίως να υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις νέες πραγματικότητες. Και αν θέλουμε στα σοβαρά να ισχυριζόμαστε ότι δεν δουλεύουμε μόνο για μας αλλά και τον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να σκεφτούμε και θέματα δημοκρατίας συμμετοχής του κόσμου. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει το έργο μας εδώ και νομίζω ότι υπάρχουν καλά επιχειρήματα για να ταχθούμε υπέρ μιας πιο μακράς περίοδου επταετούς. Και να μην αφήσουμε τους Δήμους και τις κοινότητες ε, να βρεθούν αντιμέτωπες με μια κατάσταση όπου ουσιαστικά ε, κάνουμε, ανακαλύπτουμε, μάλλον αλλάζουμε την κατάσταση κάθε πέντε χρόνια. Γιατί ήδη πολλές φορές ακούσαμε σήμερα την παράταση κατά δύο έτη του δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό γιατί θεωρώ ότι όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν ε, θα υπάρχουν ως νομική βάση γιατί θα έχουν ολοκληρωθεί. Άρα οι περιφέρειες θα πρέπει να κοιτάξουν εκ νέων τι ισχύει για τα δύο αυτά χρόνια και επί δύο χρόνια δηλαδή θεωρούν ότι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο σε δύο χρόνια θα είναι πιο πρόθυμο το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και δεν έχουμε καμία ιδέα για το πώς θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να ταχτούμε υπέρ των περιφερειών. Να ολοκληρωθεί το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο με τις... Ε, όσα έχουμε ψηφίσει. Τάσομαι λοιπόν σαφώς υπέρ των 7 ετών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος Κάρα στην αρχή. Ασχολούμαστε σήμερα με την διάρκεια των επόμενων δημοσιονομικών προπτικών, ενώ η Κομισιόν δεν είχε κάνει ακόμα καμία συνεδρίαση για να μελετήσει το πρώτο τμήμα αυτού που ε, είναι ο τίτλος της συνεδρίασής μας, δηλαδή προκλήσεις πολιτικής. Και άρα το δεύτερο τμήμα του δημοσιονομικού πόρου να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το βρίσκω αυτό πραγματικά αστείο. Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει στην άλλη αίθουσα, εδώ λίγο πιο πέρα, στα κτίρια μας. Δεχόμαστε ότι για λόγους ε, δημοσιονομικής λιτότητας αφού δεν μας δίνουν το 1% του ΑΕΠ, ε, ε, εντάξει, το δεχόμαστε. Και αφού δεν κατεβαίνουμε κάτω από το 1%, ε, το δεχόμαστε ακόμα και για 10 χρόνια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ξέρετε, έχετε καταλάβει, ότι μέχρι το 2023, 2023 δεν θα έχουμε καθόλου προχωρήσει όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Ευρώπης σε σχέση με τις πολιτικές που δεχόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τις θέσει ε, εφαρμογή μέσα στα επόμενα 13 χρόνια. Μάθανε το πιο γελίο πράγμα στο οποίο έχω συμμετέχει, είτε στην πολιτική είτε και αλλού. Εντάξει, χρειάζεται η συζήτηση για την διάρκεια των ε, δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά για όνομα του Θεού ας ασχοληθούμε με το τι θα πρέπει να καλύψουν οι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Βλέπω εδώ πέρα στο πρόγραμμα εργασία. λέει, τον Ιανουάριο θα ασχοληθούμε με τη Γεωργία. Εντάξει. Θα ασχοληθούμε με τη συνοχή και την αλληλεγγύη. Άλλο 30%. Θα ασχοληθούμε με την έρευνα και την ε, καινοτομία, ενέργεια, και διευρωπαϊκά δίκτυα, ήδη πάμε κάπως καλύτερα και έπειτα τι λέει, κάτι νέο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα νέα όργανα ελέγχου ε, δημοσιονομικού. Γιατί αν δεν ελέγξουμε δεν θα γίνει και τίποτα. Μετά λέει μεταρρύθμιση του χρηματοδοτικού συστήματος στις 28 Φεβρουαρίου και μετά ασχολούμαστε με την έκθεση. Άρα λοιπόν ένα θέμα που θα μπορούσε να απαιτήσει περισσότερη χρηματοδότηση ε, στο μέλλον, μια ψηλοσυνεδρίαση, άντε μισή μέρα. Και έπειτα θα ασχοληθούμε με τους ίδιους πόρους ή με τους πόρους γενικότερα άλλη μισή μέρα και μετά θα φτιάξουμε την έκθεση. Ε, η θα το έχει η Επιτροπή μας δεν έχει κάνει όλα, εκτός από το να μιλήσει για τις πολιτικές προκλήσεις. Και θα έχει συμφωνήσει για τη συνέχιση των δημοσιονομικών προοπτικών όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ήθελα να το πω αυτό γιατί πραγματικά με ενοχλεί από την αρχή των εργασιών αυτής της Επιτροπής. Και από δημοσιονομικής άποψης, επειδή πρέπει να το συζητήσουμε, Έχω κάποιες σοβαρές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω πώς είναι οι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν με τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς μέχρι στιγμής. Εγώ το έχω κάνει εδώ και για αρκετά χρόνια. Και σας λέω ότι ένας ε, δημοσιονομικός προϋπολογισμός για 10 χρόνια είναι το πιο γελίο πράγμα που έχω ποτέ ακούσει να προγραμματίσει κανείς για πέντε χρόνια είναι δύνατον. Για 7 χρόνια είναι δυνατόν μόνο αν έχουμε ένα άρθρο όπως αυτό που έχουμε στην υπέροχή μας συνθήκη που μας ορίζει ένα ανώτατο όριο για το τι μπορούμε να έχουμε ως πόρους και άρα και ως δαπάνες. Αυτό είναι πιο, εύκολο. Αλλά για ένα σοβαρό προπολογισμό ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί μια λογική φιλοδοξία του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ξεκινά από μια τέτοια επιτροπή σαν τη δική μας, είναι τόσο αδύνατον όσο και ένας προγραμματισμός για 10 χρόνια. Απομένει λοιπόν για να είμαστε στο ελάχιστο σοβαροί προγραμματισμός ο πενταετής. Και πάλι τι νόημα θα είχε κάτι τέτοιο. Θα είχε νόημα να μας πούνε έχουμε τη στρατηγική 2020. Από το 2013 αυτό σημαίνει στην ουσία τι, άλλα 6 χρόνια ή άλλα 7 χρόνια. Δική μου λογική κατάληξη θα ήταν ότι μέχρι το 2020 θέλουμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Από το 2013 μέχρι το 2020 έχουμε 6-7 χρόνια. Άρα οι επόμενε δημοσιονομικές προοπτικές αυτή την περίοδο θα πρέπει να καλύψουν. Και μετά από αυτόν τον προγραμματισμό θα πρέπει να έχουμε φτάσει τους στόχους που έχουμε πολιτικώς ορίσει με τη στρατηγική. Είναι το μόνο λογικό πράγμα. Αν το κάνουμε, δεν ξέρω σε τι χρησιμεύουν οι επόμενε δημοσιονομικές προοπτικέ, εκτός από το να παγιώσει ότι η Ευρώπη δεν θα δαπανίσει πάνω από το 1% του ΑΕΠ. Και φοβούμε ότι μέσα στο θεσμικό μήλο στον οποίο βρισκόμαστε είναι το μόνο πράγμα στο οποίο λογικά θα ε, χρησιμεύσουν. Θα μείνουμε σε αυτή τη μάχη την δημοσιονομική που ολοκληρώνεται τώρα και θα καλυφθούμε για τα επόμενα δύο χρόνια και στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική τα κράτη-μέλη θα μπορούν να κερδίσουν τα άλλα θεσμικά όργανα και θα πούνε οι Ευρωπαίοι δεν θα δαπανίσουν πάνω από 1% του ΕΠ. Εγώ αυτό όλα δεν τα βλέπω σοβαρά. Και ο ενθουσιασμός μου είναι σχετικά περιορισμένος και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Φυσικά, φυσικά και αντιλαμβάνομαι το σχόλιο σας. Και θα ήθελα να πω προς όλους ε, εδώ ότι το νόημα μιας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής ε, Ενό μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού δεν αφισβητείται. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε κάνει για θέματα δημοσιονομικά σε εθνικό επίπεδο, γιατί ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός σε εθνικό επίπεδο είναι θέμα Υπουργείων, Υπουργείων ε, Οικονομικών. Και αν αυτό δεν αρκεί, γίνεται ένας νέος προγραμματισμός. Στη δική μας περίπτωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Πρόκειται για μια νομοθετική δραστηριότητα και αυτό προσφέρει κάποια εχέγγυα. Γιατί το 80% του προϋπολογισμού οφείλεται σε επιχορηγήσεις. και αυτό δίνει ασφάλεια στις περιοχές και στα κράτη-μέλη. Έχω κάποιες δυσκολίες ακούγοντας ε, τις επικρίσεις εις βάρος του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού 5, 7 ή 10 χρόνια προκειμένου να υπάρχει και κάποια βεβαιότητα σε αυτό το τον προγραμματισμό και επίσης κοιτώντα τι γίνεται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο χρηματοδοτήσαμε τελικά αυτά τα οποία από ευρωπαϊκή άποψη θέλαμε να χρηματοδοτήσουμε στα κράτη-μέλη για όλους τους πολίτες. Και αυτό νομίζω ότι έχει την αξία του. James Ellis. Uh, uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως είναι θεμητό να έχουμε μια πέμπτη επιλογή για τα επτά χρόνια, γιατί αυτό έχουμε κάνει και τις τελευταίες τρεις φορές όπως αναφέρει και ο Σαλβαδόρα στο έγγραφο προβληματισμού. Αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι στο υπαριθμόν 1-2010 στα έγγραφα του ε, λεκτικού συνεδρίου που θέλουμε τη δήλωση ε, ε, ασφάλειας, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν στη διορθωτικά ταμεία. Και άρα λοιπόν δεν έχουμε τέτοια δήλωση Άρα λοιπόν ε, και στη χώρα μου όλοι λένε πως δεν ε, υπάρχει ασφάλεια στα λογιστικά της Ένωσης. Εδώ και 15 χρόνια προσπαθούμε να έχουμε αυτή τη δήλωση. Αυτά που θέλω να πω βασικά αφορούν τη δική μου εμπειρία γιατί είμαι στην Επιτροπή Προπολογισμού από το 1984. Είχαμε μια πενταετή περίοδο 84 με 89, οπότε ήταν υπέροχη περίοδο. Δεν είχαμε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Μπορούσαμε όντω να διαπραγματευτούμε έναν αδερτήσιο προπολογισμό που είχε ο καθένα τη δική του φύση. Είχαμε μάλιστα και τρει αναγνώσει μια φορά. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, στα 20 τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μείωση στη δυνατότητα τη Επιτροπή Προπολογισμού και του Κοινοβουλίου να, κρατη... να... να ασκήσει δημοσιονομικό έλεγχο. Και αυτό είναι γιατί έχουμε πολυετή προγράμματα που απομακρύνει αυτό την ευθύνη των ε, ερετών εκπροσώπων και το τοποθετεί στα χέρια των γραφειοκρατών. Νομίζω λοιπόν ότι η καλύτερη εκδοχή που μπορούμε να έχουμε είναι η υπαριθμό 3. Διότι συμφωνώ με αυτού του συναδέλφους που είπαν ότι αν επιλέξουμε το 4 και έχουμε 5 συν 5, η εμπειρία μας όχι μόνο από αυτήν εδώ την αναθεώρηση, αλλά και από την προηγούμενη που δεν έγινε καν, Βέβαια έχουμε αριθμούς, είναι δεσμευτικά στις δημοσιονομικές προοπτικές και σύμφωνα με τις συνθήκες Λισαβόνας κάθε ένας από αυτούς τους αριθμούς είναι χρυσός κανόνας όσον αφορά την εφαρμογή από πλευρά των κρατών μελών. Δεν υπάρχει ευελιξία σε μια αναθεώρηση με δεκαετή προοπτική. Αν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το δημοκρατικό έλεγχο θα πρέπει αυτό να το κάνουμε μέσω, της, μέσω του δικού μας Προεδρίου. Ο Μπαρόζο δεν έχει έλεγχο στη, δεν επηρέασε τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Τις πρώτες τις έφτιαξε ο πρώτη και μετά τίποτα. Ε, δεν είχε καμία επιρροή στο χρηματοδοτικό σύστημα γιατί ούτω ή άλλω αυτά είχαν ε, δεσμευτεί από τι δημοσιονομικέ προοπτικές και νομίζω πολύ λογικό, όπω είπαν και οι περισσότεροι συνάδελφοι, πω χρειάζεται να υιοθετήσει κανεί και να εξασφαλίσει ότι αυτή η δημοσιονομική προοπτική θα ξεκινήσει ένα μόνιμο σύστημα όπου θα έχει εκλογέ για το Ευρωκοινοβούλιο εκστρατεία εγκαίρως, όπου τα πολιτικά κόμματα θα έχουν του υποψήφιου του, θα έχουν πρόγραμμα, θα το στηρίξουν το πρόγραμμα αυτό και συμφωνώ ότι δεν χρειάζεται πάνω από ένα χρόνο για τη διαπραγμάτευση των δημοσιονομική προοπτική. Είναι σχετικά απλό. Αν έρθει η Κομισιόν και η Κομισιόν ξέρει πολύ καλά ποια προγράμματα θα θέλει να εφαρμόσει, γιατί τα έγγραφα ούτω ή άλλω έχουν συνταχθεί από την γραφειοκρατία. Και άρα έχω την εντύπωση ότι οτιδήποτε μα επιτρέπει να μπορούμε να έχουμε εκλογέ, να έχουμε προγράμματα, να λαμβάνουμε αποφάσει και έπειτα να τα εφαρμόζουμε όλα αυτά σύμφωνα με τα προγράμματα που ήδη έχουν ξεκινήσει, Νομίζω πως αυτό θα αυξήσει το δημοκρατικό έλεγχο του συστήματος και επίσης θα πρέπει να αυξήσει και την ευελιξία του. Διότι αν έχουμε ένα πενταετές πρόγραμμα θα εξασφαλίσουμε ακόμα και αν όπως είπε ο Μαρκάρα, θα έχει μέσα μια αναθεώρηση που μπορεί και να μην είναι σημαντική πάντως θα φροντίσουμε να, να ελέγχουμε τους μηχανισμούς εφαρμογής των πολιτικών. Και τελευταία μου παρατήρηση, μπορεί και ιδανική κατάσταση δεν υπάρχει στον προπολογισμό. Υπάρχουν πολλά προγράμματα ε, τα δημοσιονομ... οι δημοσιονομικές προοπτικές έχει ο καθένας το δικό του χρονοδιάγραμμα γιατί να μην σκεφτούμε και ναι, ίσως εκεί χρειάζεται για τη συνοχή περισσότερη... περισσότερα χρόνια να έχουμε για το Ταμείο Συνοχής ένα δεκαετές πρόγραμμα μόνο 5 συν 5 ναι, με αναθεώρηση στη μέση ώστε να έχουμε ένα σωστό πλαίσιο το οποίο δεν θα αποφασίζεται για όλους τους άλλους αλλά μόνο για το Ταμείο συνοχή ή να έχουμε ένα, και να έχουμε ένα γενικό πλαίσιο πενταετέ, για το οποίο είμαστε ανέκαθεν υπέρ και να κάνουμε κάτι ειδικό για το Ταμείο συνοχή που όντω χρειάζεται πιο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Πρόεδρε, να πω επίση ε, ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και από ψήφισμα στην Ολομέλεια πριν από τον Ιούνιο του επόμενου χρόνου. Γιατί διαφορετικά η Κομισιόν θα έχει ήδη αποφασίσει. Άμα περιμένουμε μέχρι τις 8 Ιουνίου για να ψηφίσουμε, θα είναι άχρηστο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το Φεβρουάριο. Μάρτιο θα πρέπει κανονικά να ψηφίσουμε, αφού θα έχουμε κάνει άλλη μια συνεδρία. Ξέρετε ότι θα έχουμε όλε τι απόψει μα, αλλά πρέπει να γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια ώστε να σφραγίσουμε αυτό που θα θέλαμε εμεί ω δημοσιονομικέ προοπτικέ, ώστε να υπάρξει δηλαδή δημοσιονομική πειθαρχία και ευελιξία ταυτόχρονα στο σύστημα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Τζέιμ, Και τώρα ο κ. Μαρινέσκο έχει το λόγο. Σας <clears throat> ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον Σαλβαντόρ για το έγγραφό του και για τον τρόπο με τον οποίο έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης. Νομίζω μας διευκόλυνε πολύ στη διεξαγωγή της συζήτησης στην Επιτροπή. Και αυτή η σωστή μεθοδολογία έχει καταλήξει σε πολύ επικοδομητική συζήτηση και σε, στη διαγραφή κάποιων απαντήσεων στις ε, ερωτήσεις. Η διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα γιατί από αυτό εξαρτάται και η κατάρτιση των περιφερειακών και των εθνικών προϋπολογισμών. Ο εθνικός προϋπολογισμός, από ό,τι ξέρω, έχει τετραετή διάρκεια. Οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα να έχουμε πιο παρατεταμένη περίοδο εφαρμογής. Στις χώρες μέλη επιλέξαμε την τετραετία γιατί αυτή είναι η διάρκεια της ε, θητείας μιας κυβέρνησης. Αλλά η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική. Βέβαια, αν είχαμε βραχύτερε δημοσιονομικέ προοπτικέ, θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε καλύτερα στι ε, αλλαγέ και στι νέε οικονομικέ συνθήκε. Αντίθετα, είναι πιο παρατεταμένη διάρκεια, μπορούμε με πιο σταθερό τρόπο να προγραμματίσουμε τα διάφορα προγράμματα. Ε, υπάρχουν δηλαδή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στι δύο απόψει. υπέρ τη βραχίας ή πιο της πιο παρατεταμένη διάρκεια. Θα πρέπει να βρούμε κάπου τη χρυσή τομή τη μέση λύση. Αν επιλέξουμε την πενταετία, όντω θα έχουμε σύμπτωση με τι θητείε τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου, αλλά θα έχουμε πρόβλημα με τι διαπραγματεύσει. Δηλαδή, μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, μετά τη σύσταση και τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από εκεί και πέρα αρχίζουμε την διαπραγμάτευση για τον προπολογισμό. Αν τα καταφέρουμε μέσα σε ένα εξάμεινο, πολύ ωραία. Αλλά μέσα σε ένα εξάμεινο το πολύ να αποφασίσουμε για τη νέα επιτροπή, για τη νέα σύσταση. Η επταετία από την άλλη πλευρά έχει δείξει ότι είναι ένα έγκυρο διάστημα, έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η πρόταση 5 συν 5, δεδομένων των συνθήκων που διανύουμε σήμερα θα ήταν η ιδεώδης λύση. Γιατί είναι ένας συνδυασμός ουσιαστικά των δύο προτάσεων. Έχουμε μία αφενός μακρά περίοδο, αρκετά μακρά για να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και εφαρμογή προγραμμάτων με μακροχρόνιο σχεδιασμό και από την άλλη πλευρά μπορούμε να προβούμε και σε ενδιάμεση δημοσιονομική διόρθωση. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα φανεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται την υποχρεωτική ρήτρα γιατί την ενδιαφέρει να εφαρμόσει όλα αυτά τα προγράμματα. Αυτή η πρόταση λοιπόν 5 συν 5 είναι κατά τη γνώμη μου η ιδανική λύση. Ε, Σας ευχαριστώ. Είναι πάντα πολύ γοητευτικό να βλέπουμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό στην χρηματοοικονομική κρίση. Αλλά και εδώ πρέπει να σας πω ότι είμαι αρκετά επιφυλακτική. Γιατί, γιατί πολύ απλά από πλευρά των κρατών μελών ε, τι ακούμε ότι είναι κακή η οικονομική κατάσταση, άρα να περικόψουμε τις δαπάνες μας, τις ευρωπαϊκές από πλευράς δικής μας θα θέλαμε να πούμε το εξή ότι αν είμαστε πραγματικά πεπισμένοι ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να γεννηθεί μέσα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. θα πρέπει να δίνουμε πιο πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια, πιο μεγάλο πιο προπολογισμό ευρωπαϊκό να έχουμε, ιδιαίτερα επειδή έχουμε την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν σε κάποιες περιπτώσεις να σκεφτόμαστε και να έχουμε ορίσει τι δημοσιονομικέ προοπτικέ και το δημοσιονομικό πλαίσιο ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ράιν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την σαφείς λύσει που μας δίνει. Είναι σημαντικό που συγκρίνουμε τις διάφορες θητείες και το δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά ακούσαμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα επίπεδο, το επίπεδο της εφαρμογής στα κράτη-μέλη ή στους Δήμους. Και να μην ξεχνάμε ότι μετά από κάθε δημοσιονομικό πλαίσιο, μετά από κάθε απόφαση για τον προϋπολογισμό, υπάρχει ένα διάστημα μέχρι να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να το λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα κοιτώντα την ε, λύση 3, η οποία μου φαίνεται λογική. Θα ήταν σωστό να σκεφτούμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Ε, αν θα ληφθεί υπόψη και για την εφαρμογή, για παράδειγμα, των 5 ετών ή αν θα πρέπει να υπάρχει και η λύση των 10 ετών σε περίπτωση που χρειάζεται για να υπάρχει και σταθερότητα. Γιατί ναι, μεν θέλουμε διαφάνεια και ε, ευελιξία, αλλά χρειαζόμαστε και στις μικρές κοινότητες ασφάλεια σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και γι' αυτό λοιπόν στον τομέα αυτό ίσως από πλευράς περιεχομένου θα είχε νόημα να υπάρχουν 10 έτη δημοσιονομικού πλαισίου. Άρα ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια, ένα συνδυασμό, να πούμε δηλαδή ότι σε κάποιους τομείς θέλουμε ευελιξία και γι' αυτό θα έχουμε πέντε έτη και σε άλλους τομείς χρειαζόμαστε σταθερότητα, άρα χρειαζόμαστε 10 έτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Η δική μου παρέμβαση θα είναι πάρα πολύ σύντομη γιατί μόλις υπόθηκαν αυτό που θέλω να πω κι εγώ. Εγώ θέλω μόνο να συμπληρώσω ένα σημείο που είναι το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Νομίζω ότι για πολλούς συμπολίτες μας η Ευρώπη υποφέρει από νομιμότητα, από δημοκρατική νομιμότητα. Πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε. Εμείς ανανεωνόμαστε κάθε πέντε χρόνια, όπως και η Κομισιόν. Είναι θεμητό η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο που κάθε φορά παίρνουν μια ανατολή θα πρέπει να εφαρμόσουν μια πολιτική, έναν προπολογισμό για τον οποίο δεν είχαν λόγο. Αυτό σημαίνει για μένα πως δεν είναι δυνατόν ο η δημοσιονομική περίοδος να ξεκινά ένα, δύο, τρεις μήνες μετά από την εκλογή του Κοινοβουλίου ή την εγκαθίδρυση νέα επιτροπή. Γιατί οι προεκλογικέ εκστρατείες τι οποίε ε, προβαίνουμε στι ε, κάστοτε χώρε μα και που βασίζονται ωραία ένα και περισσότερο σε ένα πρόγραμμα του κόμματό μα που ορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζονται σε προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά επικυρώνουν οι πολίτε και έπειτα πρέπει να τα μεταφράσουμε σε προπολογισμό. Άρα πρέπει να έχουμε ένα χρόνο για να μπορούμε να συζητήσουμε τον προπολογισμό λοιπόν, επόμενο προπολογισμό θα πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον το 2016. Δεν υπάρχει ζήτημα να ξεκινήσει το 2014, γιατί διαφορετικά η δημοκρατική νομιμότητα δεν θα μπορέσει να εκφραστεί. Και έπειτα, μέσα σε αυτή την έλλειψη νομιμότητας της οποίας είμαστε αντικείμενο, ένα τμήμα αυτού οφείλεται σε δυσκολία να ενώσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές γιατί με περιοδικό τρόπο κάθε 7 χρόνια δηλαδή αμφισβητούμε τα πάντα, τον προπολογισμό και τις διάφορες δράσεις. Ε, δεν αφήνουμε, δεν επιτρέπουμε στην κοινή γνώμη να μας παρακολουθήσει. Ας δούμε τι συμβαίνει συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια, ένα προγραμματισμό που έγινε το 2007. Τα περισσότερα κράτη χρειάστηκαν το 2008 και 2009 για να ξεκινήσουν αυτές τις νέες πολιτικές. Είμαστε στο 2010, στα τέλη του 2010 και ήδη μιλάμε για μεταρρυθμίσεις και επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές ε, δεν ξέρω πώς γίνεται στις δικές σας ε, εκλογικέ περιφέρειες, αλλά όταν εγώ επιστρέφω σπίτι μου κάθε Σαββατοκύριακο, οι άνθρωποι μου λένε «Μα, εδώ μιλάτε ήδη για μεταρρυθμίσεις, ενώ δεν έχουμε ακόμα καλά-καλά καταλάβει γιατί λάβατε την τάδε ή δίνα απόφαση στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο». Μια πολύ σύντομη λοιπόν προγραμματική περίοδο όταν είναι κακή για την νομιμότητα των πολιτικών μας και για την ε, κατανόησή τους από τους πολίτες, εκτός και αν κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη δημοσιονομική περίοδο και έπειτα την προγραμματισμό των ε, μέσων. Και γι' αυτό και συμφωνώ μετά όσο είπε η προηγούμενη ολομιλήτρια, ότι δηλαδή για τα εργαλεία, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα να ζουν περισσότερο χρόνο και να αναθεωρούμε πιο τακτικά τον προπολογισμό για να λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική πραγματικότητα. Όντω, το 2010 βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο τελείω διαφορετικό από αυτό κατά το οποίο συζητήθηκε και αποφασίστηκε αυτή η δημοσιονομική προοπτική. 5 συν 5 λοιπόν μου φαίνεται ότι είναι αποδεκτό, εάν αυτό μα επιτρέψει να προβλέπουμε ένα μια ε, αναπροσαρμογή πενταετή του προϋπολογισμού μας. Jetzt, Mr. Ουτζίας. Κύριος Ουτζίας, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω πως μετά από τη γενική συζήτηση που κάναμε μέχρι σήμερα, ο εισηγητής μας επαναφέρει στα πιο ε, πρακτικά προβλήματα σε σχέση με τα διάφορα θέματα που έχουμε συζητήσει. Άρα πιστεύω λοιπόν πως ε, είναι σκόπιμο και μετά από τη συζήτηση που έγινε σήμερα να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε λοιπόν τις θέσεις που εκδηλώνονται ανάμεσα στις διάφορες ομάδες. Έπειτα θα πρέπει επίσης να δούμε τα όρια που μας επιβάλλει η συνθήκη που προκύπτουν σαφέστατα και έπειτα και τη θέση των κρατών και του Συμβουλίου που αρχίζει να φτάνει και ως εμάς. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σίγουρα ε, την εξή έννοια, που κάτι που προέκυψε σε φέστατο, ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ε, μία ρήξη, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην αρχή του προγραμματισμού και την αρχή της πολιτικής ευθύνης όσων ε, υλοποιούν αυτόν τον προγραμματισμό. Και αυτό μας φέρνει, έτσι όπως είπε και ανέφερε και η, πως είναι η θέση της, ε, του Άλντε, όπως το ανέφερε και ο συνάδελφος Άλβαρο, μας οδηγεί στο να πούμε ότι η μοναδική θέση είναι η πενταετία. Πενταετία. Πρέπει αυτό το όριο να το λάβουμε υπόψη. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως υπάρχουν και κάποιες προβλέψεις πιο μακροχρόνιες οι οποίες δεν μπορούν να περιοριστούν στην πενταετία. Εμείς λοιπόν ως Άλντε είμαστε υπέρ της πενταετίας αλλά θεωρούμε πως πρέπει να γίνει μια μελέτη για να εμβαθύνουμε αν για ορισμένα θέματα όπως έλεγε και η συνάδελφη Ρέμερς μπορούν να αποσυνδεθούν και να προβλεφθούν με δεκαετή ορίζοντα. Εγώ πιστεύω λοιπόν και ρωτάω τον, τον εισηγητή Γκαρίγκα Πολιέντο. Ε, μπορούμε να σκεφτούμε τέσσερις βασικούς άξονες τους οποίους ε, θα μπορούν να αναγνωρίσουν όχι μόνο ένα κοινοβούλιο σε μια πενταετία, δηλαδή ε, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, οι μεγάλοι άξονες ε, διαμεθοριακών μεταφορών που δεν ολοκληρώνονται με μια έντολη, με μια θητεία. Είναι ευθύνη πολιτικών γενεών διαδοχικών και διαδοχικών πληθυσμών στις διάφορες περιφέρειες. Και να φανταστούμε λοιπόν τέτοιους άξονες οι οποίοι να, γίνονται, να προγραμματίζονται με δεκαετή ορίζοντα με δεσμευτική αρχή ότι ενδεχόμενες ε, ε, αλλαγές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν μόνο μέσω αυτών των αξώνων ώστε να μην γίνουν λιγμοί ε, μικρού καμποτάζ. Ε, θα ήθελα λοιπόν στα τελικά του σχόλια ο εισηγητή μα να μα δώσει την εντύπωσή του. σω να είναι η προσωπική του εντύπωση αυτή τη στιγμή και να επιφυλαχθεί να κάνει πιο ει βάθο παρατηρήσει αργότερα για μια τέτοιου είδου προοπτική. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Jetzt Kinga bitte. Kinga Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, προγραμματίζουμε με το μέλλον μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε και το παρόν. Δεν έχουμε ακόμη συμφωνία για τον προπολογισμό του 2011. Ευελπιστούμε ότι θα συνάψουμε συμφωνία σύντομα, αλλά είναι δύσκολο να διαπραγματευτούμε δημοσιονομικά θέματα με το Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται. Λέμε ότι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη στη διάρκεια της κρίσης και το Συμβούλιο λέει ναι μεν, αλλά δεν έχουμε πόρους για την επόμενη περίοδο. Οπότε η κρίση δεν διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις, ούτε διευκολύνει την ε, παγίωση κάποιων ε, μακροχρόνιων προοπτικών ή τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό. Πάντως, διαπιστώνουμε ότι τα κριτήριά μας δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν μερικές φορές. Οπότε δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμη οι διοργανικές σχέσεις και το πλαίσιό τους. Ευελπιστούμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στο μέλλον και θα είναι πιο εύκολη η σύναψη συμφωνιών. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υλοποιήσει ένα τέτοιο στόχο. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε τώρα δεν είναι να έχουμε περισσότερο χρόνο για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Υπάρχει και άλλο θέμα. Υπάρχει το θέμα της δημοκρατικής νομοποίησης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποια αποθεματικά σε κάθε δημοσιονομική γραμμή, ώστε και το σημερινό κοινοβούλιο αλλά και τα επόμενα να μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους χωρίς να υπονομεύουν τη σταθερότητα του προϋπολογισμού. Και φυσικά χρειαζόμαστε και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Γιατί έχουμε την πολιτική συνοχή, στην γεωρική πολιτική. Τέτοιες πολιτικές χρήζουν μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Βέβαια όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με τους σπόρους που έχουμε στη διάθεσή μας όσο λιγότερα κονδύλια έχουμε, τόσο περισσότερες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε για να εφαρμόσουμε τις ε, πολιτικές μας. Οπότε κατά τη συζήτηση της διάρκειας, δεν ξέρω αν θα αυτή θα είναι πενταετής, επταετής ή δεκαετής, να βρούμε και έναν άλλο τρόπο για την κατανομή των κονδυλίων, γιατί το μέχρι τώρα σύστημα δεν λειτουργήσε πολύ εύρυθμα. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε και αρκετούς δημοσιονομικούς πόρους για τις νέες πολιτικές. Δεν βλέπω τόσο τεράστιες διαφορές μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών διαδικασιών και της ευρωπαϊκής ε, διαδικασίας για τον προϋπολογισμό. Φυσικά δεν μπορούμε να αλλάζουμε τον προϋπολογισμό μας κάθε χρόνο, αλλά υπάρχουν ε, στοιχεία του προϋπολογισμού που θα μπορούσαν κάλλιστα να αναθεωρούνται κάθε χρόνο. Αν έχουμε μία επταετή διάρκεια, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε αποθεματικά που θα μπορούν να υπάγονται σε διετή αναθεώρηση, ώστε να έχουμε εξασφαλίσει και τη λογοδοσία και την διαφάνεια και τη σταθερότητα. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Κίνγα αναφέρθηκε στην σταθεροποίηση των διαθεσμικών σχέσεων και ότι δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα ουσιαστικά μετά τη Λισαβόνα. Δεν ξέρω. Άκουσαμε και μια χοροδία. Δεν ξέρω αν ήταν κάποια συγκεκριμένη ένδειξη αυτή. Τέλο πάντων, Καταρίν. Ο κύριο Ιβάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο που μέχρι στιγμής ε, δεν το ακούσαμε ιδιαίτερα. Μιλούμε για την ελαστικότητα και τη σταθερότητα αλλά να μην ξεχνούμε και την αποτελεσματικότητα. Γιατί μιλούμε για την έγκριση του προπολογισμού των, των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών κτλ. Αλλά η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα και πολύ αργή εξαιτία τη απροθυμία και τη κολυσιεργία των κρατών μελών. Αν θέλουμε πιο αποτελεσματικού μηχανισμού, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρώτα απ' όλα χρόνος. Και κάθε νέα πολιτική που θα εφαρμόζουμε θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύστημα ελέγχου και εφαρμογής των κοινοτικών κονδυλίων. Σε μία πενταετία δεν προλαβαίνουμε να εφαρμόσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη εξαιτία των ιδιαιτεροτήτων τους και των ειδικών προβλημάτων τους τα διάφορα προγράμματα. Είναι πολύ στενή αυτή η περίοδο. και δεν έχουμε μόνο τις νέε χώρε που αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά και τις ε, παλιότερε. Στην πολιτική συνοχή προβλήματα υπάρχουν σε πολλές χώρες, σε παλιές και σε νέες. Οπότε θα πρέπει να είμαστε με φιλόδοξοι και να είμαστε διορατικοί, στραμμένοι προς το μέλλον, γιατί έχουμε πια πολύ, πολλές προκλήσεις ε, καινούριε. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Ίσως η καλύτερη πρόταση είναι αυτή του 5 συν 5 με μια ισχυρή ρήτρα ενδιάμεση αναθεώρησης. Νομίζω ότι αυτή είναι η ιδανική λύση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ja, vielen σας ευχαριστώ και αν δεν υπάρχει κανένας άλλος που θέλει το λόγο, θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κάνει μια πρώτη σύνοψη και να κάνει τα πρώτα του σχόλια σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έγινε. Και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το εξής. Καταρχάς, πώς τοποθετείται ο συνάδελφος στις προτάσεις των συναδέλφων που προτείνουν κάποια πολιτικά ζητήματα, κάποιοι πολιτικοί τομές να μην ε, προσαρμόζονται στο δημοσιονομικό πλαίσιο, να αφαιρεθούν από το δημοσιονομικό πλαίσιο και να τους δοθεί ε, μεγαλύτερη προθεσμία. Η πολιτική συνοχή, τα τένς, τα... Ε, οι μεταφορές διεθνικές, η έρευνα και αντομία, δεν ξέρω αν θα έρχεσαν και αυτά σε αυτό τον τομέα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Να υπάρχει ένα διαχωρισμός δηλαδή μεταξύ των μέσων και των γενικών δημοσιονομικών προοπτικών. Και το δεύτερο θέμα που θέλω να ακούσω είναι σε ό,τι αφορά τις εργασίες της Επιτροπής μας. Η ιδέα του James που λέει ότι, ότι το Μάρτιο θα έπρεπε να κάνουμε ίσως μία ενδιάμεση συζήτηση για να δώσουμε και να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα όσα έχουμε αποφασίσει ενδεχομένω ω τότε στην Ολομέλεια και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου. Σάλβα, τώρα έχεις το λόγο. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακούσαμε πολλές ενδιαφέρουσες και εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά και ποικίλε. Γιατί δεν ακούσαμε ούτε δύο πανομοιότυπες απόψεις σχεδόν σε όλη αυτή τη συζήτηση. Κάτι που καθιστά τις συνεισφορές πολύ πλούσιες και καρποφόρες και δυσκολεύω βέβαια τον εισηγητή, γιατί δημιουργήθηκε ένα ψηφιδωτό προτάσεων και απόψεων που δίνει μία αίσθηση της πολυφωνίας της Επιτροπής μας, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το μέλλον των δημοσιονομικών προοπτικών. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο σας σχόλιο, με την πιθανότητα δηλαδή θέσπισης διαφορετικών περιόδων προγραμματισμού άλλων συντομότερων και άλλων πιο παρατεταμένων. Δεν έχω αντίρρηση, απλώς έχω την αίσθηση ότι αυτό θα πρέπει να το σχεδιάσουμε στα πλαίσια των εγκάρσιων πολιτικών που θα εξετάσουμε μεταγενέστερα, για παράδειγμα την πολιτική συνοχής ή την γεωργική πολιτική πρώτα απ' όλα. αυτή την άποψη η περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να είναι πιο μακροχρόνιες. Ο κύριος Σουτζίες μίλησε για τις υποδομές μεταφορών, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, για την έρευνα. Οπότε επανερχόμαστε στην αρχική ιδέα του εισηγητού, που προέβη σε μία συνολική ανάλυση, γιατί οι περισσότερες προτεραιότητες περιλαμβάνονται στη στρατηγική του 2020 και άρα είναι λογικό η διάρθρωση των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών να συνδυάζεται με την στρατηγική του 2020. Όπως ακούσαμε και από πολλούς ομιλητές που παρουσίασαν διάφορες ιδέες. Η δική μου ιδέα ήταν τα πέντε χρόνια. Και εγώ προτίμησα την πενταετία γιατί έχω πολύ πολύχρονη πείρα στην Επιτροπή Προπολογισμών. Και όπω και άλλοι συνάδελφοι που παρακολούθησαν για πολλά χρόνια τι εργασίε τη Επιτροπή Προπολογισμών, έχουν αυτή την εμπειρία τη δυσκολία. Ε, ε, ελαστικότητα σε εθνικούς προϋπολογισμούς, σε αιτήσεις προϋπολογισμούς, όταν έχουμε ανελαστικές δομές δημοσιονομικών προοπτικών. Και η επταετία ήταν αρκετά ανελαστική. Δεν εξασφαλίζει αυτή την ευελιξία που χρειαζόμαστε για, τις αιτήσεις, για τους αιτήσους προϋπολογισμούς. Και πολλές φορές προσκρούσαμε σε εμπόδια στην εφαρμογή των πολιτικών μας γιατί δεν υπήρχε κανένα περιθώριο, καμία δυνατότητα ελαστικής εφαρμογής του προϋπολογισμού. Επιμείναμε πολύ σε αυτό το θέμα της ελαστικότητας και η ελαστικότητα των τελευταίων δημοσιονομικών προοπτικών οφείλεται ακριβώς στην ε, χαμηλή εφαρμογή της δεύτερης κατηγορίας που είναι η κοινή γεωρική πολιτική. Και αυτό δεν το προτιμάει κανένας, ούτε η υπέρμαχη της κοινή γεωρικής πολιτικής, ούτε τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Κάποιος που ασχολείται, που είναι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ίσως θέλει πιο σύντομη βραχία διάρκεια δημοσιονομικών προοπτικών. ενώ ε, συνάδελφοι όπως η κυρία Κρέλη, που είναι μέλος της ε, Επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυξης, κάποιος που είναι μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, για παράδειγμα, θα προτιμούν πιο μακροχρόνιες περιόδους προγραμματισμού. Η εναλλακτική λύση του 5 συν 5 είναι πολύ επικίνδυνη και το επισήμαναν ο κύριος Πόρτας και ο κύριος Άσουαρθ γιατί 5 συν 5 δεν σημαίνει δύο φορές 5. Η εναλλακτική λύση 5 συν 5 ουσιαστικά ακυρώνει, εξουδετερώνει οποιαδήποτε δυνατότητα ελαστικής χρήσης του προϋπολογισμού, γιατί προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια κάθε κατηγορίας και θα ήταν πολύ δύσκολο, εκτός και αν φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς υποβάλλουμε μια πολύ πρωτότυπη πρόταση ενδιάμεσα αναθεώρησης. Αλλιώς ξεχάστε την ελαστικότητα στον προϋπολογισμό με την πρόταση 5-5. Γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει τα ανώτατα όρια της δεκαετίας ανώτατα όρια που θα είναι τελείω ε, αμετάκλητα ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια τη περίοδου. Εκτό κι αν, επαναλαμβάνω, έχουμε μια πολύ ειδική ρήτρα ενδιάμεση αναθεώρηση και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανεί να διανοηθεί τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια τέτοια ρήτρα ενδιάμεση αναθεώρηση για να μα εξασφαλίσει μια ελαστικότητα. Οπότε θα είχαμε μονίμω δυσφορία καθ' όλη τη διάρκεια τη δεκαετία. Επταετία. Η επταετία εξακολουθεί να είναι μια έγκυρη εναλλακτική λύση. Θα μπορούσαμε και αυτή να τη συμπεριλάβουμε στο έγγραφο, αλλά αυτή ήδη ισχύει τώρα. Αλλά και στην προηγούμενη, στις δύο προηγούμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές είχαμε ε, παραπονεθεί για την ανελαστικότητα αυτής της επταετούς διάρκειας. Οπότε θα προτιμούσαμε μία ρήτρα πενταετία. Αυτή τουλάχιστον είναι η γνώμη του εισηγητού. Φυσικά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις τομεακές πολιτικές, την πολιτική συνοχή, πολιτική, τη γεωργική πολιτική και να επανέλθουμε. Πάντως και η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχή. αν ε, συντομεύσουμε τους ε, χρόνους διάρκειας θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και την πολιτική συνοχής και ως προς την εφαρμογή τις συμβάσεις εκτέλεσης. Χρειαζόμαστε και γραφειοκρατική διοικητική απλούστευση, γιατί στο έγγραφο μιλήσαμε για απλούστευση και βελτίωση στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Στη γεωρική πολιτική επίσης είναι προφανές ότι για τον προγραμματισμό προτιμούμε μια πολύ πιο παρατεταμένη περίοδο προγραμματισμού, αλλά είμαι βέβαιος ότι με τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής που εγκαινιάστηκε από τον Επίτροπο Σόρος θα, θα μπορούσαμε να βρούμε λύση και σε συντομότερες δημοσιονομικές προοπτικές. Και η πρόταση παράτασης κατά μία διετία των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών προκειμένου να περάσουμε αργότερα στην πενταετία αυτό δεν θα πρέπει να το εξετάσουμε ως λύση εργασίας, αλλά ως έκτακτη λύση σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας. Στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές, η διαπραγμάτευση δεν έγινε σε περίοδο κρίσης, αλλά σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. Το 2005 και το 2006 δεν είχαμε την τωρινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Και είχαμε προεδρίες βαρέων βαρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Τόνι Μπλερ, τη Βρετανική Προεδρία, τον Γιούνκερ στην Προεδρία του Λουξεμβούργου, τον Καγκελάριο ε, που ολοκλήρωσε ε, εκ μέρους Αυστριακής Προεδρίας ε, τις δημοσιονομικές προοπτικές. Χρειάστηκαν τρεις προεδρίες και 18 ολόκληροι μήνες για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Και ήταν μια πολύ θετική στιγμή επαρχιών Αγελάδων. Δεν νομίζω το Συμβούλιο ότι είναι σε θέση ούτε τώρα ούτε το 2011 να επισέλθει σε μια εις βάθος συζήτηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Και πολύ δύσκολο θα ήταν το Συμβούλιο σε θέση το 2013 να καταλήξει σε δημοσιονομική συμφωνία με 27 χώρες μέλη. Η τρίτη εναλλακτική λύση είναι αυτή που προτιμάτε φαίνεται γιατί είναι η μόνη που μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε σε πενταετή περίοδο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε ένα facing in, μια σταδιακή εφαρμογή για την πενταετή περίοδο. Πάντως συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για πενταετίες αν δεν λάβουμε προηγουμένως υπόψη τις ανάγκες των τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των γεωργικών πολιτικών, όπως της γεωργικής πολιτικής, της ε, πολιτικής συνοχής, πολιτικής έρευνας, αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυρία Πρόεδρε. Πολλοί συνάδελφοι έφυγαν δυστυχώς και έτσι δεν θα απαντήσω στις επιμέρους παρατηρήσεις, αλλά θα λάβω όλα αυτά τα σχόλια ως βάση για το έγγραφο εργασίας. Τώρα, ως προς το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την εκπόνηση ενός εγγράφου που θα μπορούσαμε να υποβάλουμε το Φεβρουάριο ή Μάρτιο προς την Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι αρκεί η συζήτηση για το έγγραφο. Θα πρέπει να στηριχθούμε στο γεγονός ότι για την Ολομέλεια θα εγκρίνουμε έγγραφο τον Ιούνιο. Φυσικά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και feedback από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το 5 συν 5, που κατά τη γνώμη μου δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε με μια σαφή πρόταση που δεν θα χρήζει κατά ανάγκη εγγράφου, αλλά μιας πολιτικής συζήτησης και μιας αποκριστάλλωσης πολιτικής γνώμης εκ μέρους της Επιτροπής. Πάντως, ελπίζω και η δική μας συζήτηση να επηρεάσει τις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε είναι χρέος του εισηγητού, του συντονιστού, της Προέδρου να έχουμε σταθερές ε, και τακτικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρχει μεγάλη απόκληση στις προτάσεις. Αυτά κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες των προτάσεων που ακούσαμε. Λαμβάνω υπόψη όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις για, ως βάση για τις μελλοντικές για τα μελλοντικά έγγραφα εργασία και νομίζω ότι έγινε μια πολύ καρποφόρα και πλούσια συζήτηση. Πάντως όλοι συμφωνούμε ότι χωρίς μεγαλύτερη ελαστικότητα του προπολογισμού, ο μηχανισμός του κοινοτικού προπολογισμού δεν πρόκειται να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στις πολιτικές προκλήσεις που μας επισήμανε ο κύριος Έγγελς. Έφυγε βέβαια στο μεταξύ, αλλά θα ήθελα να απαντήσω και σε αυτή του την μορφή. Εμείς καταρτήσαμε ένα πλαίσιο εργασίας στο οποίο προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε συνένεση και για να βρεθεί πολιτική συνένεση το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι μια τεχνική βάση. Αρκετά στέρη που είναι καρπός μακροχρόνιας συζήτησης και αυτή είναι η προϋπόθεση πριν περάσουμε στη συζήτηση για τις πραγματικές πολιτικές που είναι και οι πολιτικές ε, προκλήσεις, αλλά χωρίς τεχνική βάση και χωρίς συγκέντρωση μιας συμφωνίας δεν μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη φάση. Αυτό το νόημα είχε και η εντολή της Επιτροπής ΣΟΥΡ να διαμορφώσει αυτή την τεχνική βάση. Και μετά θα επισέλθουμε στα πιο επιμάχα θέματα για τις μεταρρυθμίσεις των κοινωτικών πολιτικών και τι χρειάζεται ε, για να ανταποκριθούμε σε αυτές με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ. Αναμένουμε λοιπόν το έγγραφο εργασίας, τα έγγραφα εργασίας μάλλον, τα οποία θα μας υποβάλλει ο εισήγητης και θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα τα έχουμε στη διάθεσή μας. Ζητά κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Έχουμε ακόμα χρόνο στη διάθεσή μας και αν στο 4, στα διάφορα δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα συνάδελφος που να ζητάει το λόγο, στο σημείο αυτό κλείνει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας και είμαι πεπισμένη γιατί πολλές φορές θα συναντηθώ με όλους τους συναδέλφους και την επόμενη εβδομάδα, αλλά επειδή στην παρούσα σύνθεση ε, συνεδριάζουμε για τελευταία φορά στο τρέχον έτος. Σας εύχομαι και σε εσά και στις οικογένειές σας καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, να επανέλθετε σόι και αυλαβείς υγιής καρτιμελής τον Ιανουάριο και θα τα ξαναπούμε από το νέο έτος. Καλό βράδυ.